71 in commissione. Ora, oh, Cari colleghi, è un piacere riprendere. Con συνάδελφοι, e χαρά. Συνεχίζουμε. La τις δραστηριότητες στη συνάντηση με την Προεδρία του Συμβουλίου. Ευχαριστώ τον Υπουργό Γκαλέτη. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τον Ιταλό Υπουργό <clears throat> Περιβάλλοντος, πολύ ιδιαίτερη, γιατί αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη μετακίνηση του Κώστα Κονκόρδια θα ήθελε να είναι στη γέφυρα του Κροαζιεροπλίου, το οποίο θα εγκαταλείπει επιτέλους το ωραίο νησί του Τζίλιο Παρ' όλα αυτά προτίμησε να έρθει εδώ και θα του δώσω το λόγο αμέσως για να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας για το επόμενο εξάμεινο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο confronto e soprattutto per darmi l'opportunità di illustrarvi e di Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα το περιβαλλοντικό της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. subito di sottolineare una cosa, la volontà di questa presidenza η επιθυμία μας είναι να συνεργαστούμε με συνεχή και αποτελεσματικό τρόπο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ορισμένες λύσεις θετικές ε, που δεν θα είναι δυνατόν ίσως να τις να τα κλείσουμε αυτά τα θέματα ε, και επίσης να ακούσω και τις απόψεις και σε άλλα θέματα τα οποία εσείς θα μου υποδείξετε επιμένω σε αυτό. Αν πράγματι θέλουμε αυτό το εξάμεινο να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά και κατά τη διάρκεια εσείς της εντολής σας να δουλέψετε αποτελεσματικά η στενή συνεργασία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι θεμελιώδης. Έχω την αίσθηση ότι για τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, για τα θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος. Δεν μπορούν να υπάρχουν μόνο ε, διαφορές. Δεν μπορεί να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Στόχος μας είναι να βρούμε μία συμφωνία για να λύσουμε προβλήματα τα οποία είναι ευρωπαϊκά, είναι εθνικά, αλλά είναι και παγκόσμια. Το πρόγραμμα για το περιβάλλον λοιπόν εμπνέεται από τα θέματα επίσης της ανάπτυξης και της πράσινης απασχόλησης και ε, λαμβάνει υπόψη και την ε, κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά από τις συναντήσεις κορυφής ή μάλλον τις συναντήσεις ε, του Συμβουλίου για το Περιβάλλον κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής και της Ελληνικής Προεδρίας, τις οποίες ευχαριστούμε για την πολύ καλή τους δουλειά. Λοιπόν, ανάπτυξη και απασχόληση. Εμείς ιδιαίτερα στο περιβάλλον μπορούμε στα πλαίσια του ορισμού του συγκεκριμένου στόχου να πετύχουμε κάτι το πολύ θετικό. Πρόκειται για μια πολιτιστική ανατροπή. Να θέσουμε το περιβάλλον στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Να προστατεύσουμε βέβαια το περιβάλλον γιατί αυτός παραμένει ο αρχικός μας στόχος, αλλά ταυτόχρονα να δείξουμε ότι στην Ευρώπη, στις χώρες μας και στον κόσμο δεν θα πρέπει να υπάρξει ε, μια μία υφόρος ανάπτυξη και δεν θα υπάρξουν νέες θέσεις απασχόλησης αν το περιβάλλον δεν είναι η βασική μας ανησυχία είναι καθοριστικό για το μέλλον, για την ανάπτυξη και αυτή είναι η πολιτιστική ανατροπή την οποία πρέπει να κάνουμε. Και σήμερα για να το πετύχουμε μας υποστηρίζουν και τα δεδομένα. Αν υπάρχει ένας τομέας ο οποίος κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης συνέχισε να αναπτύσσεται και σε επίπεδο κύκλου εργασιών και σε επίπεδο απασχόλησης είναι η λεγόμενη πράσινη οικονομία. Επί τη βάση λοιπόν αυτής της διαπίστωσης θα πρέπει να κάνουμε ένα περαιτέρω πολιτισμικό άλμα και να δείξουμε σε όλους στην Ευρώπη πώς. η ανάπτυξη και η απασχόληση μπορεί να γίνουν όχι μόνο μέσα και ε, διαμέσου της πράσινης οικονομίας αλλά και στους υπόλοιπους οικονομικούς τομείς ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι ε, θεωρούνται οι πιο επιθετικοί για το περιβάλλον. Τσιμεντοβιομηχανία ένα ναι. παράδειγμα. Εκεί το περιβάλλον πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πρέπει να μην αγνοηθεί η πράσινη οικονομία αλλά να μην μείνουμε και μόνο στην πράσινη οικονομία. Το περιβάλλον θα πρέπει να διαχυθεί σε όλους τους τομείς της παραγωγής. Η Ιταλική Προεδρία επανειλημμένα έχει υπογραμμίσει ότι η προτεραιότητά μας είναι η <clears throat> ανάπτυξη και η απασχόληση. Αν θέλουμε να οδηγηθούμε στην ανάκαμψη και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη ε, στους Ευρωπαίους για την Ευρώπη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Το τελευταίες εκλογές μας έστειλαν ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Αν δεν είμαστε σε θέση να πάρουμε γρήγορες αποφάσεις προς το συμφέρον και εξυπηρετώντας τους πολίτες που εκπροσωπούμε, όχι μόνο εμείς δεν θα μείνουμε στην ιστορία, αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύουμε να βυθίσουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αν δεν το προσπαθήσουμε. Απαιτείται λοιπόν η ανατροπή. Οι πολιτικές οι περιβαλλοντικές είναι πολιτικές που στηρίζουν οι κοινέ γνώμες όλων των χωρών και είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για να συγχρονίσουμε εκ νέου τις πολιτικές με τις επιθυμίες των πολιτών. Η οικονομική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών, είναι όλα αυτά για την Ιταλική Προεδρία, τμήμα της σωστή στρατιστικής. Είμαστε πεπισμένοι ότι η ανάπτυξη την οποία πρέπει να επιδιώξουμε, αυτή η οποία θα συνδυάσει το περιβάλλον με την παραγωγικότητα, είναι η πράσινη οικονομία. Στο Μιλάνο, στην ανεπίσημη συνάντηση που είχε γίνει ανάμεσα στις Επιτροπές ε, Εργασίας και Περιβάλλοντος, πριν μερικούς μήνες συναντήθηκαν όλοι οι Υπουργοί Περιβάλλοντος με όλους τους Υπουργούς Εργασίας σε μια ενιαία συνάντηση για να συζητήσουν τι μέσα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χώρες μας για να μπορέσουμε εμείς να αντισταθούμε στην πανόλη που χτυπά την Ήπειρό μας, δηλαδή την ανεργία και ιδιαίτερα την ανεργία των νέων. Η επιτυχία της συνάντησης αυτής του Μιλάνου δείχνει ότι κάτι τέτοιο πρέπει να συμβεί για να αυξήσει τις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης έτσι ώστε να περάσουμε σε μια οικονομία χαμηλής παραγωγής διοξιδίου του άνθρακα και που θα βασίζεται σε αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων και πηγών κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα προσπαθήσουμε και μέσα από το έγγραφο για την ανάπτυξη το οποίο σημειώνει αν θέλετε την έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να αναφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο στα θέματα της πράσινης οικονομίας. Είναι ένα θα έλεγα μήνυμα για το ότι η οικονομική διακυβέρνηση της ζώνης ευρώ λαμβάνει υπόψη την πράσινη οικονομία. Θα προτείνουμε εμείς να μην συμμετείχουν στις προσπάθειες αυτές ε, οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Υπουργοί Εργασίας αλλά και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος για να ληφθούν πάντα υπόψη από τους υπόλοιπους ε, τα θέματα του περιβάλλοντος. Όπως κάθε σημαντική μεταρρύθμιση και αυτή από την κρίζα οικονομία δηλαδή στην πράσινη οικονομία θα έχει και πιθανώς κάποιες αρνητικές συνέπειες σε μία πρώτη φάση. Κάποιες κατάλληλες λοιπόν κοινωνικές πολιτικές πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες των αλλαγών στην βιομηχανική πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 Αντιπροσωπεύει λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία έτσι ώστε η περιβαλλοντική διάσταση να ληφθεί υπόψη στη διαδικασία της οικονομικής διακυβέρνησης. Η επιλογή μας είναι να ανατρέψουμε και να ξεπεράσουμε με αποφασιστικό τρόπο την παραδοσιακή εικόνα της σχέσης οικονομικών πολιτικών και περιβάλλοντος που πολλές φορές ε, εκ των υστέρων μόνο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες σε περιβαλλοντικό επίπεδο των οικονομικών πολιτικών. Οι οικονομικές επιλογές δεν θα πρέπει να μην λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις γιατί οι εμπειρίες μας πλέον μας δείχνουν ότι ο σεβασμός του περιβάλλοντος και οι αξίες του σεβασμού του περιβάλλοντος είναι τόσο βαθιά αγκυρωμένες στην Ευρώπη που είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη από τη βιομηχανία. Είναι καθήκον λοιπόν και των βιομηχάνων να κάνουν στρατηγικές επιλογές που σέβονται το περιβάλλον και αυτό θα μας επιτρέψει και θα τους επιτρέψει να μεγιστοποιήσουν και τα κέρδη τους. Είναι λοιπόν και αυτό μια απόρρεια της πολιτιστικής αλλαγής που απαιτείται. Να πετάξουμε λοιπόν, να δημιουργήσουμε τις βάσεις για μια κυκλική οικονομία που θα καλύπτει τις ανάγκες, όχι να μένουμε στο παίρνω, μετατρέπω και μεταπετάω. Μιλάμε για ε, ειδική αξίας πρώτες ύλες, παράγοντας όμως τελικά εν πολλή απόβλητα, σκουπίδια. Αυτό το πρότυπο είναι απαράδεκτο, είναι κάτι που μολύνει, δημιουργεί κρίσεις και κατά συνέπεια δημιουργεί απώλεια θέσεων απασχόλησης και φυσικά και απώλεια κέρδους για τους βιομηχάνους. Στα πλαίσια της συζήτησης που έγινε στο Μιλάνο φάνηκε ότι πρέπει να ενισχύσουμε την περιβαλλοντική διάσταση της οικονομικής governance της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο περιβάλλοντος και σε επίπεδο διαδικασιών. Ως Προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος λοιπόν κατά τη διάρκεια των επομένων μηνών θα προσπαθήσω να δημιουργήσω το σωστό περιβάλλον για να συμπεριληφθεί η περιβαλλοντική διάσταση στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μετά από τις συστάσεις της ανεπίσημης συνάντησης του Μιλάνου η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντική. Εύχομαι λοιπόν να μπορέσει να βγει από τις συζητήσεις σας θετικά στοιχεία προς την κατεύθυνση αυτή. Είμαι πεπισμένος πως τα βασικά θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τα μη αναβαλώμενα πλέον, ε, οι, οι αποφάσεις που δεν μπορεί πλέον να αναβληθούν από εδώ και πέρα θα βοηθήσουν να συνδυάσουμε τις πολιτικές μας προσπάθειες και έτσι θα μπορέσουμε εμείς να καθοδηγηθούμε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να είμαστε παρόντες εδώ. Δεν θα πρέπει εμείς ε, απέναντι σε κράτη που κάνουν ακατανόητα βήματα προς τα πίσω να μείνουμε αδρανείς. Πάρα πολύ συχνά η Ευρώπη ε, επιβραδύνει την ανάπτυξή της από τοπικισμούς και από απαράδεκτες επιλογές. Η Ιταλική Προεδρία λοιπόν θέλει ε, στον τομέα του νομοθετικού πλαισίου να ορίσει τα πράγματα σωστά και στο κλίμα και στην ενέργεια. Θα υπάρξει λοιπόν με ένας οδικός χάρτης, με κάποιες ανεπίσημες συζητήσεις. Αντιμετωπίσαμε στα πλαίσια του Ανεπίσημου Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος και το θέμα της ανταλλαγής εκπομπών και προβλέπεται να ξανασυζητήσουμε στο Ανεπίσημο Συμβούλιο Ενέργειας στις 6 Οκτωβρίου ε, τα θέματα αυτά, ιδιαίτερα τα θέματα της ενέργειας. Είμαστε πεπισμένοι ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των κλιματολογικών άλλαγων συνδέεται με την διασφάλιση της προμήθειας ενέργειας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προετοιμάσουμε και τη συνάντηση κορυφής για το κλίμα στη Λίμα του ΟΗΕ ε, ήδη παρουσιάσαμε τις πρώτες θέσεις μας στη Βαρσοβία από τον προηγούμενο χρόνο έτσι ώστε να καταλήξουμε στις τελικές εθνικές συνεισφορές για την Ισφαιρική Συμφωνία του 2015. Αυτά θα οδηγήσουν στη διάσκεψη του Παρισίου τον επόμενο χρόνο που θα είναι η κρίσιμη στιγμή για όλους. Η συνάντηση των ηγετών κορυφής του Ban ki θα είναι μια ευκαιρία έτσι ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε, ε, για την προετοιμασία της συνάντησης των Παρισίων το 2015. Εγώ θα ήθελα να είναι παρούσες όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ακουστούν οι συνεισφορές τους και οι προτάσεις τους. Αγαπητά μέλη λοιπόν, η Ιταλική Προεδρία θα ε, συνεχίσει στην συνάντηση του Συμβουλίου στις 28 Οκτωβρίου και στις 17 Δεκεμβρίου του 2014, σύμφωνα πάντα και με τις τυπικές προθεσμίες, κάποιες διαδικασίες και κάποιες αποφάσεις σε θέματα σημαντικά. Απαιτείται λοιπόν για να το πετύχουμε η στενή συνεργασία μαζί σας. Στον τομέα των περιβαλλοντικών το θέμα των γενετικά τροποποιημένων είναι η βασική προτεραιότητα νομοθετική της Προεδρίας. Μετά από πολλά αίτια δράνεια, στασιμότητα στις 12 Ιουνίου καταλήξαμε σε μια πολιτική συμφωνία η θέση του Συμβουλίου έχει σαν στόχο μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση του συστήματος αδειοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απέτηση από πλευρά των κρατών μελών να περιορίσουν τον, την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων στο έδαφος τους και να το ορίσουν ανάλογα με τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά τους. Έναν τομέα τόσο ευαίσθητο, ο οποίος εμπλέκει το σύνολο της κοινωνίας, από τους γεωργούς, τους καταναλωτές, θα πρέπει να αναγνωριστούν τα επίπεδα αυτονομίας και κυριαρχίας των μεμονωμένων κρατών μελών. Η κοινή γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει στείλει τα σωστά μηνύματα και, τον τρόπο και για τον λόγο αυτό είναι πολιτικό μας καθήκον να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν σε μια συμφωνία ανάμεσα σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Σήμερα το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ε, ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Βασική μας ευχή λοιπόν είναι να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε εγκαίρως να κλείσουμε τη συμφωνία με, για τα γενετικά τροποποιημένα. Το επόμενο θέμα είναι η μείωση της χρήσης ε, σε πλαστικές σακούλες. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει όχι απλά να μειώσουμε τις ποσότητες των πλαστικών σάκων που χρησιμοποιούμε, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια ευκαιρία για τη βελτίωση του συνολικού ε, πακέτου διαχείρισης αποβλήτων. Απαιτείται μια συμφωνία η οποία θα μας επιτρέψει να λάβουμε υπόψη μας τις ισχύουσες διατάξεις και τις ε, χρηστές πρακτικές οι οποίες ήδη υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Εύχομαι λοιπόν ότι η κυρία Άουκεν θα μπορέσει να αποκτήσει μια σωστή διαπραγματευτική εντολή τον Σεπτέμβριο δημιουργώντας εσύ τις βασικές προϋποθέσεις για να καταλήξουμε σε μια γρήγορη συμφωνία. Τώρα για τη μείωση των εκπομπών σε αέρια θερμοκηπίου. Το πρόγραμμα το νομοθετικό της Προεδρίας προσανατολίζεται στην ολοκλήρωση των ρυθμίσεων που έχουν ήδη περάσει. Η πρόταση κανονισμού για την παρακολούθηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών είναι βασική μας προτεραιότητα. Η οδηγία επίσης για τη χρήση της γης, η λεγόμενη οδηγία μας ε, ε, έχει απασχολήσει πολύ. Πρόκειται για ένα θέμα δύσκολο, μια διαπραγμάτευση δύσκολη και η πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ενέργειας στις 13 Ιουνίου αντικατοπτρίζει τις δύσκολες ισορροπίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Συνειδητοποιούμε ότι, στο κοινοβούλιο, αυτή, ε, ότι το Κοινοβούλιο έχει προτείνει μια διαφορετική οδό οι προτάσεις του κυρίου Τόρβαλτς είναι μια πρόταση η οποία θα διασφαλίσουν μια συμφωνία όμως με το Συμβούλιο. Η πρόταση επίσης για την απόφαση τη σχετική με τον μηχανισμό ελέγχου των αερίων είναι κάτι το θετικό. Υπάρχει επίσης και το θέμα του ETS. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να σταθεροποιήσουμε το θέμα του ETS στα πλαίσια της καταπολέμησης ε, των κλιματολογικών αλλαγών γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε το χρόνο αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε τις ε, κύριες διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό, αλλά ελπίζουμε να βάλουμε τις βάσεις για μια γρήγορη ε, προώθηση του θέματος. Υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα, πρόκειται για σημαντικότατες προτάσεις, οι οποίες είναι τμήμα αναπόσπεστο μιας μακροπρόθεσμης και ισχυρής περιβαλλοντικής πολιτικής. Περιμένοντας λοιπόν από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκεκριμένες θέσεις, εμείς θα προωθήσουμε το ταχύτερο δυνατόν τις εργασίες μας στο Συμβούλιο, κάνοντας μια εξέταση σε βάθος των προτάσεών σας. Η Ιταλία Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συντονίσει και θα καταθέσει τις θέσεις της Ένωσης και στα διεθνή φόρα. Ανάμεσα στις διεθνείς αυτές συναντήσεις θα σας θυμίσω ορισμένες. Καταρχάς η διάσκεψη του τμήματος της Σύμβασης για τη βιολογική πολυπλοκότητα και ταυτόχρονα ε, και οι συναντήσεις ε, των χωρών που έχουν υπογράψει τα πρωτόκολλα της Καρταχένα και της Ναγκόγια. Ε, θα υπάρξει η συνάντηση COP12 η οποία θα γίνει στη Νότια Κορέα στα, στις, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Εκεί θα αποφασιστούν οι περαιτέρω δράσεις που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της κατάστασης και την επίτευξη των στόχων του ΆΙΚΙ. Αλλά ταυτόχρονα επίσης θα υπάρξει και η προσπάθεια αναδιατύπωσης των στόχων στα πλαίσια της προσπάθειας των Ηνωμένων Εθνών η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίξει έναν ρόλο επικοδομητικό εφαρμόζοντας πλήρως τις αποφάσεις των προηγουμένων διασκέψεων. Θα ήθελα να κλείσω ευχαριστώντας σας για την προσοχή σας. Θα ήθελα επίσης να σας εμπιστευθώ ότι σε θέματα όπως όλα αυτά τα οποία άπτονται του περιβάλλοντος και με τα οποία εσείς ασχολείστε, και εμείς στο Συμβούλιο και εσείς στην Επιτροπή σας μπορούμε να συνεργαστούμε στενά με επικοδομητικό τρόπο και χωρίς προκαταλήψεις. Το περιβάλλον και το θυμίζω για μια ακόμη φορά περισσότερο από πάρα πολλά άλλα θέματα άπτεται της ζωής και του μέλλοντος όχι μόνο ημών των ιδίων αλλά και των επομένων γενεών. Καλές δουλειές κύριε Πρόεδρε Λαβία και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ για την τόσο λεπτομερή παρουσίασή σας της, ε, του προγράμματος της Ιταλικής Προεδρίας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μέσω ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων, δίνοντας το λόγο στους συντονιστές, τους οποίους παρακαλώ όμως να περιοριστούν σε δύο λεπτά για τις παρεμβάσει τους και θα υπάρξει μετά μια πρώτη απάντηση από την πλευρά του κυρίου, ε, του κυρίου Γκαλιέτη. Έχει το λόγο καταρχήν ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Εγώ Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία ως συνοριστής του ΕΛΚ να υποδεχτώ δύο υπουργούς από την Ιταλική Προεδρία, οι οποίοι ανήκουν και οι στο ΕΛΚ. Η Ιταλική κυβέρνηση δεν είναι μόνο μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών και χαίρομαι για την παρουσία σας κύριε Υπουργέ επειδή έχετε θέσει ως προτεραιότητά σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το σημαντικό γεγονός της μετακίνησης του Κώστα Κονκόρδια το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητά σας. Εγώ επανέρχομαι στις δηλώσεις σας για το στόχο του 2030, 2030. Είναι απαραίτητο να πράξουμε τα απαραίτητα ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο να μπορέσει να δεχτεί μια πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο ΕΛΚ φυσικά. Δεν υπήρξε καμία διαφωνία για το θέμα αυτό γιατί μίλησα με τους συναδέλφους μου να μπορέσουμε να θεσπίσουμε αυτό το στόχο του 40% ο οποίος είναι αδιαμφισβήτητος για εμάς. Και ζητούμε λοιπόν να τον δεχτεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Φυσικά υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ακόμα και στο κόμμα μου μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το αν θέλουμε να έχουμε ένα ή τρεις στόχους. Αλλά η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και η πλειοψηφία της ομάδας εργασίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος θεώρησε ότι πρέπει να θεσπίσουμε τρεις στόχους γιατί βάσει της ε, ίδιας της έκθεσης αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θεωρούμε ότι αυτό θα είναι καλύτερο, θα ενισχύσει το δυναμικό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με την τεχνολογία περιβάλλοντος. Πιστεύω λοιπόν ότι σήμερα είχαμε μια πολύ σημαντική απόφαση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι 30% η αύξηση ενεργειακής απόδοσης μέσα στο πακέτο αυτό. Ελπίζω λοιπόν ότι τουλάχιστον αυτό θα γίνει δεκτό από το Συμβούλιο και θα υπάρξει υποχρεωτικός χαρακτήρας, θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για το περιβάλλον και θέλω να τονίσω ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων σε μια στιγμή που είναι τεταμένες οι σχέσεις μας με τη Ρωσία, ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο τη βιομηχανία μας να αποκτήσει μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Δίνω το λόγο τώρα στο Ματιό Γκρότα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ, χαίρομαι που θέλετε να προωθήσετε μια πολιτιστική στροφή, η βιομηχανία να περάσει σε ένα πιο αηφόρο τρόπο και να υπάρξει ένα θετικό ανταγωνισμό, ο οποίο θα δημιουργήσει θέσει απασχόληση και θα τι εξασφαλίσει στον τομέα του περιβάλλοντο. Πολλοί συνάδελφοι εδώ έχουν παρουσιάσει ιδέε για τα θέματα αυτά, για το πώ θα μπορούσαμε να προωθήσουμε την εργασία μας σε σχέση με το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Και φυσικά για το σύνολο της περιβαλλοντικής ε, ε, νομοθεσίας. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε αυτή την σταθερότητα με τον Ιβο το οποίο ήταν ο εισηγητής μας και να έχουμε μια σταθερή άποψη. Ε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το 2021 το οποίο προτείνει η Κομισιόν είναι πολύ καθυστερημένο Φοβάμαι ότι το σύστημα το ETS θα έχει ήδη υποστεί μεγάλες ζημίες και θα είναι πολύ έργα για την τροποποίησή του. Γι' αυτό θέλω να προτάξω το 2017 ως έτος εφαρμογής των αλλαγών. Για την διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή, την διάσκεψη COP. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρούσα σε αυτές τις συνεδριάσεις με την Επιτροπή, φυσικά συνοδευόμενη από μία αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου <clears throat> και η Κομισιόν είναι πάντα έτοιμη να δράσει, αλλά πολλές φορές φαίνεται ότι υπάρχουν 28 διαφορετικές εθνικές απόψεις οι οποίες αναδύονται. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η Ιταλική Προεδρία να μπορέσει να εξασφαλίσει μια κάποια ενότητα, ιδίω για τα θέματα χρηματοδότηση όπου δεν υπάρχει πάντα συμφωνία μεταξύ των κρατών μέλων. Για το θέμα τη ενεργειακή απόδοση. Είναι κάτι το οποίο είναι περισσότερο αυτό το οποίο πετύχαμε, περισσότερο από αυτό το οποίο ελπίζαμε, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε περισσότερα. Μεταξύ του 40 και του 30% υπάρχει μια διαφορά 10%. Θέλουμε να έχουμε μια αύξηση της ενεργειακής απόδοσης η οποία να είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό θα ήταν πραγματικά ένα θετικό πρόγραμμα και το οποίο θα μπορούσε σε μόνιμο επίπεδο και με αϊφόρο τρόπο να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Ελπίζω ότι η Προεδρία θα είναι ανοιχτή <clears throat> για να μπορέσουμε να έχουμε και μια πιο φιλόδοξη αντιμετώπιση και αυτό το οποίο έχει αποφασίσει η Κομισιόν να μην γραφεί στις ανάδελτους της ιστορίας και να είναι αποφασισμένο χωρίς καμιά αλλαγή. Ο Γιάννη Ντάνκεν έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Σε ολόκληρη την Ευρώπη ανησυχούμε για θέματα ασφάλειας και ενεργειακής και θα θέλαμε να ξέρουμε τη θέση του Υπουργού για την συμβατική ενέργεια που διαθέτουμε από τους υδρογονάνθρακες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα για τους φιλελεύθερους ο Νίλ Στόρβαλτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γκαλέτη για την παρουσία σας. Με μεγάλη χαρά σας ακούσαμε και ελπίζουμε να ικανοποιηθούμε και το Σεπτέμβριο όταν θα σας πούμε αριβεντέρτσι. Ακούγονται φήμες ότι στο Συμβούλιο μπορεί να υπάρξει μία μειοψηφία που θα μπλοκάρει τα πράγματα. Μπορείτε να μας πείτε τι δυνατότητες έχετε να το αντιμετωπίσετε αυτό, Μίλε Γκράτσιε. Ευχαριστούμε. Κατερίνα Κονέτσνα. Δεν ακούω. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος της GUE NGL. Ξέρω ότι το έργο σας δεν θα είναι εύκολο. Γιατί? Εμείς θα σας υποστηρίξουμε πλήρως, αλλά θα ζητήσουμε και από σας συγκεκριμένες ενέργειες. Θέλω να δεσμευτείτε ότι εσείς θα αγωνιστείτε για να υπάρξει αμέσως μια επιγραμμική διαβούλευση για την συμφωνία TTIP με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει να κάνει με το περιβάλλον αυτή η συμφωνία, έχει να κάνει με τη χημική βιομηχανία, έχει να κάνει με την ασφάλεια των τροφίμων, έχει να κάνει με μια σειρά από πρότυπα τα οποία έχουμε εγκαθιδρύσει στην Ευρώπη και φοβόμαστε ότι στις ε, διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ η Κομισιόν δεν θα τα υποστηρίξει όλα αυτά. Θα πρέπει εσείς να αναλάβετε ένα ηγετικό ρόλο και θα θέλαμε να έχουμε και από εσά διευκρινήσεις για το ποιε είναι οι προοπτικές για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Για μας, όπως φαίνεται τα πράγματα τώρα, είναι τελείως απαράδεκτα και φοβόμαστε ότι τα κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα του περιβάλλοντος είναι υποαπειλή μέσα στις διαπραγματεύσεις αυτές. Θα ήθελα επίσης να σας θέσω το ερώτημα πώς αντιμετωπίζετε το θέμα της οικονομίας των αποβλήτων. Μιλάτε για μια κρίση αποβλήτων, μιλάτε ότι όλα, για το γεγονός ότι όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Αλλά πώς μπορείτε να λύσετε αυτό το πρόβλημα στην Ιταλία. Υπάρχει μια πραγματική κρίση σε σχέση με τα απόβλητα από ό,τι γνωρίζω. Και η κρίση αυτή έχει και επιπτώσει στον υδροφόρο ορίζοντα. Πώ θα λύσετε αυτό το πρόβλημα, τι είδου πρότυπα θέλετε να εισαγάγετε, ώστε να μην υπάρχει η ρήπανση από τα απόβλητα στη χώρα Σα. Ευχαριστώ. Ο Ικχάουτ από, του πράσινου. τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό για την πλήρη παρουσίασή του του προγράμματος Ιταλικής Προεδρίας για τους επόμενους μήνες. Προβλέπετε να είναι μια μεγάλη πρόκληση και πολύ ενδιαφέρον για τους επόμενους μήνες. Όταν έλεγε ο, η συνάδελφος από τους πράσινους Αριβεντέρτσι, νομίζω ότι το έλεγε με ένα φιλικό τρόπο για να ξαναβρεθούμε μετά το καλοκαίρι. Μία από τις μεγάλες προτεραιότητες για μας βέβαια θα είναι το ενεργειακό πακέτο για το 2030 και στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ενωμένη για το θέμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμω είναι ενωμένο. Έχει μια σαφέστατη θέση για το πώ πιστεύουμε ότι το ενεργειακό πακέτο θα πρέπει να διαμορφωθεί ώστε να παραμείνει ένα πακέτο. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να έχουμε τρει δεσμευτικού στόχου. Μείωση των εκπομπών, ποσοστό των ε, ανανεώσιμων ενεργειών που να μεταφράζεται σε εθνικού στόχου και ενεργειακή απόδοση. Η Κομισιόν μόνο 30% προέκρινε το στόχο αυτό για μέχρι το 2030 παρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει 40% και είχε ζητήσει να είναι δεσμευτικό αυτό ο στόχο. Περιμένουμε λοιπόν από την Ιταλική Προεδρία να προωθήσει το Συμβούλιο προ την επίτευξη μια συμφωνία πακέτου για του τρει δεσμευτικού στόχου και θα ήθελα να ακούσω περισσότερα από τον κύριο Υπουργό για το πώ θα προωθήσει το θέμα αυτό στι συζητήσει στο Συμβούλιο. Ένα άλλο θέμα είναι η συνάντηση τη ΚΟΠ στη Λίμα, όπω αναφέρατε, και ένα από τα κύρια θέματα τα οποία θα συζητηθούν το θέμα τη χρηματοδότηση των ενεργειών για την προστασία του κλέματο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπατε, δεν έχει ποτέ μια κοινή θέση γιατί είναι τα κράτη-μέλη τα οποία δεσμεύονται για χρηματοδότηση. Και αυτό είναι κάτι το απρόβλεπτο, αστάθμητο και οδηγεί σε μια ασάφεια σε σχέση με τη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Θα μπορέσετε λοιπόν για αυτό το επόμενο μισό έτο να εξασφαλίσετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάει στη λίμα με μια ενιαία φωνή, μια ενιαία θέση για τη χρηματοδότηση και όχι μόνο αστάθμητε και αβέβαιε θέσει των κρατών μελών. Τελευταίο ερώτημα για την παρακολούθηση των εκπομπών από την Αυτό θα είναι ένα από τα σημαντικά θέματα ε, σε νομοθετικό επίπεδο που ελπίζουμε να περατώσουμε στην Ιταλική Προεδρία και ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα διαφάνειας που είναι το ελάχιστο που πρέπει να επιτύχουμε από τη δική μας άποψη. Θα μπορέσετε λοιπόν να εξασφαλίσετε μια σαφή θέση του Συμβουλίου για την διαφάνεια σε σχέση με τις εκπομπές από, θα, από σκάφη στη θάλασσα. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, ο Πιέ Νικόλα από την ομάδα του FDD. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσίασή του και να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Εγώ εκπροσωπώ εδώ ένα πείραμα γιατί όπως γνωρίζετε ανήκω στην ομάδα FDC και στο κόμμα των πέντε αστέρων και εμένουμε σε θέματα όπως η άμεση δημοκρατία και το ερώτημα που θα θέσω είναι ένα ερώτημα που πολλοί Ιταλοί πολίτες θα ήθελαν να θέσουν. Τι εννοώ. Λαμβάνοντας υπόψη τις φιλόδοξες ε, προτάσεις σας ε, για τη μείωση κατά 30% των καυσαερίων και για αύξηση κατά 30% των εναλλακτικών πηγών ενέργειας ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις οικονομικές επιπτώσεις. Πώς κρίνει λοιπόν την απόφαση που είχε πάρει η κυβέρνηση Μόντι για, την, για το διπλασιασμό της παραγωγής ε, ε, υδρογων στην Ιταλία και σε υπηρετικό επίπεδο και σε θαλάσσιες περιοχές όπως ακριβώς συμβαίνει και στην Κροατία. Τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν μπορεί να είναι και κίνδυνοι για καρκίνο και στην Ιταλία και στην Κροατία λόγω ακριβώς της δημιουργίας όλων αυτών των σημείων εξόριξης και αν πράγματι το θέμα είναι να βγάλει κανείς χρήματα δεν θα πρέπει ίσως να διπλασιάσουμε από το 7 σε 14% τον ποσοστό κέρδους του κράτους και όχι να διπλασιάσουμε την παραγωγή. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσε ο πρώτος γύρος λοιπόν των συντονιστών. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Υπουργό για να δώσει τις πρώτες απαντήσεις, όχι πάνω από πέντε λεπτά παρακαλώ αν γίνεται, γιατί είναι πολλοί συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Δύσκολο είναι, θα προσπαθήσω όμως. Σας ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη αν δεν σταθώ σε όλες τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, 30% βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτές είναι οι τελευταίες προτάσεις της Επιτροπής. Εγώ νομίζω ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει πάρα πολύ στη Συμφωνία Κλίμα Ενέργεια του 2030. Όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου, πρόκειται για ένα στρατηγικό στόχο της Προεδρίας και για το σύνολο του Συμβουλίου και το Κοινοβούλιο. Είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται πλήρως και με τους στόχους που έχουμε θέσει εμείς σαν Ιταλική Προεδρία. Είναι σαφές ότι η βελτίωση στον τομέα της αποδοτικότητας της ενέργειας δημιουργεί περισσότερο κύκλο εργασιών, μεγαλύτερο κύκλο εργασιών για τις επιχειρήσεις ε, επηρεάζει την ασφάλεια του περιβάλλοντος, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, μας επιτρέπει να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να είμαστε και περισσότερο ανεξάρτητοι στο επίπεδο της διασφάλισης πηγών ενέργειας. Πρόθεση του Συμβουλίου λοιπόν είναι να εργαστεί όσο περισσότερο γίνεται έτσι ώστε να μπορέσουμε στις 26 Οκτωβρίου να ε, καταλήξουμε σε μια συνένεση σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλουμε στους ε, Ευρωπαίους πολίτες και όχι μόνο. Ιδιαίτερα στη συνάντηση ε, της Λίμα το Δικέμβριο και στο Παρίσι το 2015. Προφανώς υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πιο ενάρετες, mm. χώρες πιο φιλόδοξες και χώρες λιγότερο φιλόδοξες. Στόχος της Ιταλικής Προεδρίας θα είναι να καταλήξουμε στην πιο φιλόδοξη δυνατή συμμαχία που θα συνδυάζει τις προσπάθειες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα για τα ETS, το είπα και στην παρουσίασή μου είναι κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με τη συμφωνία ανάμεσα στο κλίμα και στην ενέργεια. Θα πρέπει το Συμβούλιο Υπουργών να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν. Ας περιμένουμε λοιπόν. Πρέπει να πετύχουμε είναι κάτι το οποίο θα καταστήσει την αγορά πιο αξιόπιστη, θα την καταστήσει πιο διαφανή και θα μειωθούν έτσι οι εκπομπές καυσερίων. Περιμένουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει ε, σημαντικές προτάσεις, θα προσπαθήσουμε να τις λάβουμε υπόψη όταν τις ολοκληρώσετε, ελπίζω να μην καθυστερήσουμε και να συνεχίσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Για το e-look, ξέρετε ότι πάνω σε αυτό το θέμα έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία τον προηγούμενο Ιούνιο. Εμείς θέλουμε να καταλήξουμε το ταχύτερο δυνατόν με την οδηγία αυτή, με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συζήτηση δεν είναι εύκολη. Σε κανένα από τα δύο θεσμικά όργανα η συζήτηση αυτή δεν πέρασε εύκολα αλλά αυτό ακριβώς ε, μπορεί να οδηγήσει το Συμβούλιο ε, ε, να προωθήσει μια θέση που θεωρούμε ότι είναι ένας καλός συμβιβασμός. Όπως είπα λοιπόν υπάρχουν δυνατότητες για τη συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Σαν Ιταλική Προεδρία εμείς διαπραγματευόμεθα με δεκτικό πνεύμα ε, και σχολιάζουμε επίσης ε, ε, και, εξετάζουμε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου. Οι κανόνες που μας εμπνέουν είναι ο παραλληλισμός, η αμοιβαία αναγνώριση και ο σεβασμός των κοινωνικών, οικονομικών, αξιακών επιπέδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω σε αυτές τις αξίες και πάνω σε αυτά τα κριτήρια εμείς δεν θα υπαναχωρήσουμε. Θα συνεχίσουμε και θα απαιτήσουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια σχετικά με τα απόβλητα Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε ε, σημασία σε όλες τις ε, απόψεις ε, και σε όλα τα θέματα και στο θέμα των αποβλήτων. Τώρα δεν θα μπω στα θέματα που αφορούν άμεσα τη χώρα μου γιατί εγώ έχω έρθει εδώ σήμερα σαν εκπρόσωπος του Συμβουλίου και δεν θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά στα Ιταλικά θέματα αλλά υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες φτάνουν στη χώρα μου σε επίπεδα ανακύκλωσης που είναι τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Ε, εμείς δεν έχουμε το πρόβλημα των αποβλήτων οξύτερα από άλλες χώρες, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα, είναι όμως θέμα που αφορά το σύνολο της Ευρώπης. Το πακέτο για τα απόβλητα έγινε πρόσφατα δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά συνέπεια είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταστεί προτεραιότητα στη διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι σημαντικό για μας. Περιμένουμε τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στόχος μας θα είναι να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στις εργασίες του Συμβουλίου. Αυτό θα είναι μια απτή απάντηση για τη σημασία που δίνουμε στα θέματα των αποβλήτων και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα τον Οκτώβριο να συζητήσετε τις πρώτες θέσεις μας. Σχετικά τώρα με τις εκπομπές της θαλάσσιας μεταφορές. Εμείς αναγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία που έχει αυτό το θέμα και στα πλαίσια του IMO Εμείς γνωρίζουμε ε, το αποτέλεσμα της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να την εξετάσουμε περισσότερο προσεκτικά χρειαζόμαστε χρόνο. Ε, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε ε, γρήγορα στην αίτηση για συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, για την τελευταία ερώτηση είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Δεν θα ήθελα να το αντιμετωπίσω μόνο για τη χώρα μου, για την Ιταλία. Να θυμίσω ότι και στην Ιταλία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη γνωρίζουμε εμείς ποιες είναι οι συνέπειες ε, των προβλημάτων αυτών. Ποιες, τι, più restrittive in, in, in Europa, Eh, Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δώσουμε εμείς στο θέμα αυτό μεγάλο βάρος ε, και δεν θα πρέπει ε, να το αγνοήσουμε στο μέλλον. Και για το ε, σχιστολιθικό φυσικό αέριο δεν υπάρχει νομοθετικό έγγραφο ακόμα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση ε, για το, τις συνέπειες τις περιβαλλοντικές που μπορεί να έχει το σχιστολιθικό αέριο σε μια ήπειρο σαν την Ευρώπη και η Ιταλική Προεδρία θα διευκολύνει φυσικά τη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις στον πρώτο αυτό γύρο ερωτήσεων. Έχουμε άλλους 24 τώρα συναδέλφους οι οποίοι έχουν ζητήσει να λάβουν το λόγο. Θα κάνουμε μία δόση με 12 συναδέλφους και μια δεύτερη απάντηση του κύριου Υπουργού και μετά θα συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε με τον Ιβο Μπέλετ από το ΕΛΚ. Και σας λέω και πάλι δύο λεπτά το πολύ, σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να σεβαστώ αυτό το όριο. Κύριε Υπουργέ, σας χαιρετώ ξανά και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και την προθυμία σας να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Βέβαια έχουν τεθεί ήδη οι σημαντικότερες και δώσατε ήδη εξαιρετικές απαντήσεις. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή μέρα γιατί εκφράζεται σήμερα η πρόταση της Κομισιόν για το στόχο του 30% και γνωρίζουμε και συμφωνούμε όλοι ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι κάτι πολύ ζωτικό για να μειώσουμε την ενεργειακή μας εξάρτηση ως προς τη Ρωσία. 5% πιο μεγάλη μείωση. Αυτό σημαίνει 11% λιγότερη χρήση αερίου. Περιμένουμε λοιπόν τα μέσα Οκτωβρίου και υπολογίζουμε στην Ιταλική Προεδρία ώστε να, με την υποστήριξη όλων των χωρών μελών να γίνει αποδεκτός αυτός ο στόχος της ενεργειακής αποδοτικότητας. Το ερώτημά μου κύριε Πρόεδρε αφορά, κύριε Υπουργέ μάλλον, αφορά την εμπορία των πασαστώσεων. Και ο ένας συνάδελφος προηγουμένως ήδη σας μίλησε για τη διαρθρωτική αλλαγή που χρειάζεται μεταρρύθμιση. Γιατί ξέρουμε ότι έχουν μειωθεί πολύ οι τιμές, δεν υπάρχουν πια κίνητρα σχεδόν για να επενδύσει η βιομηχανία σε καινοτόμες τεχνολογίες. Ελπίζουμε λοιπόν να συμφωνείτε ότι η διαρθρωτική μεταρρύθμιση είναι κάτι απαραίτητο και ότι πρέπει να προχωρήσει το θέμα αυτό. Αυτή η πρόταση της Κομισιόν τους επόμενους μήνες γνωρίζουμε ότι βέβαια μόνο στα τέλη του χρόνου θα μπορέσει να εγκριθεί τελικά. Ελπίζω όμως μέσα στην Προεδρία σας. Ο Ματίας ήδη σας ρώτησε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτής της μεταρρύθμισης γιατί μερικές χώρες μέλη και όχι οι μικρότερες θέλουν να παρεμποδίσουν τα πράγματα. Να μην μιλήσουμε για το 2020 αλλά για το 2017 θέλουν ορισμένοι. Το υπάρχον σύστημα ποσοστώσεων θα ισχύσει μέχρι το 20, αλλά μήπως μπορείτε να μας πείτε κάτι για, προσωπικά για το χρονοδιάγραμμα που εγκρίνεται και για τις ποσοστώσεις που είχαν χορηγηθεί από πέρυσι. Backloaded. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο από την ομάδα των Σοσιαλιστών το λόγο. Κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για την προσεκτική σα και αναλυτική και παθιασμένη παρουσίαση του προγράμματο για το περιβάλλον τη Ιταλική Προεδρία και για τη διάθεσή σας να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση λοιπόν. Στα πλαίσια της αναθεώρησης της ε, οδηγίας 94-26 ε, για ε, τα απόβλητα που δημιουργούνται κυρίως από... E allora io le chiedo cosa intende fare la Presidenza su questi target, come pensa... Από τις συσκευασίες ε, πώς μπορείτε εσείς ε, να συνδυάσετε τον ευρωπαϊκό στόχο τη χρήση των ε, πλαστικών σάκων και ταυτόχρονα με κάποιες εθνικές πολιτικές οι οποίες διαφοροποιούνται όπως η Ιταλία. Στα πλαίσια της παρουσίασής σας παρουσιάσατε με πολύ συνθετικό τρόπο την αντιμετώπιση του νέου πακέτου για τα απόβλητα. Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να επιταχύνετε προς την κατεύθυνση αυτή ε, και τι ε, βήματα προόδου θα έχουν γίνει στο τέλος του εξαμήνου. Ευχαριστώ για την ομάδα των συντηρητικών η κυρία Γκίρλινγκ. My apologies, Chairman. Too busy talking. Um, Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, μιλούσα με το γειτονά μου. Ένα απλό ερώτημα σας θέσω. Κύριε Υπουργέ, κάνατε μια εισαγωγική παρουσίαση των προτεραιοτήτων σας και μεταδώσατε κατά κάποιο τρόπο ένα είδο περίληψη τη ατζέντα τη Ιταλική Προεδρία για την περιβαλλοντική πολιτική τη. Εγώ δεν κατάλαβα πολύ καλά σε τεχνικό, σε συγκεκριμένο επίπεδο, τι θα ζητήσει από τους αξιωματούχους του να προωθήσουν ως προτεραιότητα τους επόμενους μήνες. Μήπως θα μπορούσε να μα πει Ποιε είναι οι τρει πρώτε σα προτεραιότητε, ποια είναι τα τρία θέματα που θέλετε να διεκπαιρεώσετε και που θέλετε να είστε στο τέλο τη Προεδρία σα. Ευχαριστώ για την ομάδα Άλντε η κυρία Ρής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί βλέπω ότι είναι κάπως αθλητικού χαρακτήρα η άσκηση στην οποία αποδίεται ο κύριος Υπουργός. Θέλω να επανέλθω σε ορισμένα ευαίσθητα ζητήματα, παραδείγματος χάρη το θέμα των γενικά τροποποιημένων οργανισμών και την ικανότητα των κράτων, κρατών μελών να περιορίζουν την καλλιεργιά τους. Εγώ έχω ε, διοριστεί συγγήτρια για το θέμα αυτό πρόσθετα. Πρόσφατα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, υπερευαίσθητο σε ορισμένε περιοχές και παίρνει και κριτικό χαρακτήρα σε ορισμένε περιοχές. Η κοινή γνώμη δεν παρακολουθεί μονάχα με ενδιαφέρον, αλλά έχει κινητοποιηθεί οι γεωργοί και οι καταναλωτέ περιμένουν πολλά από εμά, έχουν αναποθέσει τι ελπίδε του σε εμά, είναι πολύ ψηλό ο πύχη. Μας είπατε για την κοινή θέση του Συμβουλίου ότι έχει συμφωνεί στο Συμβούλιο, Εμεί δεν την ξέρουμε ακόμα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να σα υπενθυμίσω όμω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε μια πολύ σαφή άποψη, 500 ε, ψήφοι εναντίον 80 περίπου, σχεδόν ομοφωνία, είναι πολλά πράγματα λοιπόν για τα οποία εμεί δεν θέλουμε να υποχωρήσουμε. Και η πρώτη ανάγνωση για το θέμα αυτό ανατρέχει το 2011. Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια που έχει μείνει στο ψυγείο του Συμβουλίου. Σήμερα το απόγευμα δεχτήκατε πολύ αισιοδόξω ότι κατά τη δική σα Προεδρία θα μπορέσετε να επιτύχετε θετικά αποτελέσματα ακόμα και κλείσιμο του φακέλου. Εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ να επιτευχθεί αυτό, αλλά θέλω να σα ρωτήσω τι σα κάνει να πιστεύετε κάτι τέτοιο. Ποιοι είναι οι λόγοι που σα κάνουν τόσο αισιόδοξο Ξέρω ότι μακροηγόρησα λιγάκι. Δεν θα θέσω άλλα ερωτήματα, εκτός από ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ ζωντανό <clears throat> στο Βέλγιο μεταξύ των πολιτών μας. Είναι η σπατάλη των τροφίμων. Όλοι μας έχουν ερωτήσει για τα θέματα αυτά. Είναι 90 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων που κατασπαταλώνται κάθε χρόνο, που καταλήγουν στα σκουπίδια. Είπατε ότι και αυτό το θέμα θα σας απασχολήσει κάπου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το θέμα και στην αγανάκτηση των πολιτών. Τι προβλέπετε να κάνετε για αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Άουκεν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήλθατε λοιπόν και σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι αναφερθήκατε στην έκθεσή μου για τους, τις πλαστικές σακούλες. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και ελπίζω θα θέσετε όση πίεση είναι δυνατόν να τεθεί για να τονίσετε ότι πρέπει να γίνουν πράγματα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την πρόταση που έθεσε πραγματικούς στόχους μείωσης της χρήσης των πλαστικών σάκων και όλοι μπορούσαν να τεθούν σε μία μείωση κατά 50% για 3 χρόνια και 80% σε 5 χρόνια. Και επίσης ζητήσαμε να υπάρχει ένα υποχρεωτικό σύστημα τιμολόγησης για τις πλαστικές σακούλες, τουλάχιστον για αυτές που χρησιμοποιούνται για τα τρόφιμα. Ξέρω ότι η Ιταλία έχει προχωρήσει πολύ στα θέματα αυτά με την νομοθεσία της. Ελπίζω λοιπόν θα μας υποστηρίξετε εκεί και ότι θα συνεχίσετε το έργο σας για την αντιμετώπιση των αποβλήτων και τη μείωση των αποβλήτων γιατί αυτή είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε στα σοβαρά τη μείωση των αποβλήτων με τη μείωση της ε, απόλυψης αποβλήτων και την πρόληψη των αποβλήτων και για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Θεωρούμε ότι ίσως και η επόμενη υπουργό θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, αλλά ελπίζουμε και εκεί ότι εσείς θα ακολουθήσετε τη γραμμή του κυρίου Γιούνκερ, λέγοντας ότι δεν είναι αποδεκτό όταν τα δύο τρίτα των κρατών μελών είναι εναντίον των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, να μπορούν ακόμα να καλλιεργούνται. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια λύση η οποία θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό και επανερχόμενη στα απόβλητα. Πήγα πολλές φορές στην Καμπανία με την Επιτροπή Αναφορών και στο Λάτσιο με την Επιτροπή Αναφορών. Είναι θαυμάσια μέρη αυτά στην Ιταλία που έχετε καλά συστήματα αλλά έχετε και αποτρόπια παραδείγματα που τα πράγματα πηγαίνουν πραγματικά στραβά νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να πιέσετε την Κομισιόν να λύσει τα προβλήματα αυτά και η Κομισιόν να μπορέσει να παίξει ένα πρωταρχικό ρόλο για τη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά φυσικά πρέπει να λύσετε το πρόβλημα της καμπανίας. Σας ευχαριστώ πριν δώσω το λόγο στους επόμενους ομιλητές. Παρακαλώ. Ε, υπάρχει μια αλλαγή στο πρόγραμμά μας. Ξέρω ότι θα ήταν χρήσιμο να θυμηθούμε ότι κρατήθηκε ένα λεπτό σιγής στην Ολλανδία για τα θύματα της πτήση της Μαλαισιανής. σα δώσω όλους ένα λεπτό σιγής από τη δική μας πλευρά επίσης. Grazie eh, Σας ευχαριστώ για τη συμβολική πράξη που είναι τόσο σημαντική. Δίνω το λόγο τώρα στον Μάρκο Αφρόντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, επανέρχομαι στο θέμα το οποίο θέσατε με γενικό τρόπο. Η ha messo all'asta nel mare Adriatico 29 aree in cui eh, andare eventualmente ad estrarre idrocarburi. Eh, ξέρουμε ότι στην Αδριατική υπάρχουν θέματα τα οποία μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια λόγω ακριβώς των ερευνών για πετρέλαιο ανάμεσα στην Κροατία και την Ιταλία ε, έχει προχωρήσει η Κροατία περισσότερο από ότι στην Ιταλία. Είπατε ότι υπάρχουν κάποιες οδηγίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα ε, αυστηρές. Νομίζω ότι ε, σε μια περιοχή η οποία είναι τόσο περιβαλλοντικά επιβαρημένη όπως η Αδριατική, οι πιθανότητες εξόριξης και αναζήτησης υδρογοναθράκων θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα η κυρία Γκαρντίνη. Θα είμαι σύντομη, θα περάσω στην ερώτησή μου απευθείας, σας ευχαριστώ βέβαια για την παρουσίασή σας. Να έρθω λίγο στο θέμα της διάσκεψης της Λίμα. Εγώ μέχρι την Κοπενχάγη παρακολούθησα προσεκτικά όλες τις κόπ. Τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι είδαμε την τελευταία στιγμή να ξεπερνιούνται κάποιες δυσκολίες που είχαν δημιουργηθεί και πολλές φορές ε, υπήρχαν φόβοι ότι οι διαδικασίες δεν θα κατέληγαν σε επιτυχία. Ε, με λοιπόν για την περίπτωση της συνάντησης στο Παρίσι. Τι θα συμβεί για να μην αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα συνειδητοποιούμε τη δυσκολία της κατάστασης πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση η οποία αντιπαραθέτει την ανταγωνιστικότητα με το κλίμα και την ανταγωνιστικότητα με το περιβάλλον. Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσετε λίγο περισσότερα στοιχεία και κάτι άλλο το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αναφερθήκατε στην ανεπίσημη συνάντηση του Μιλάνου ανάμεσα στους Υπουργούς Απασχόλησης και τους Υπουργούς Περιβάλλοντος. Τι θα κάνει η Ιταλική οικονομία, η Ιταλική κυβέρνηση γύρω από την λεγόμενη κυκλική οικονομία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω ένα πολύ απλό ερώτημα. Οι ενδοκρινικές ανομαλίες έχουν ε, κατεβεί στις προτεραιότητες. Η Κομισιόν δεν μας δίνει τις πληροφορίες που ζητάμε και θα ήθελα να γνωρίζω αν η Προεδρία σας που ήταν μάλλον να ε? μάλλον ασαφής για αυτό το θέμα σκοπεύει να κάνει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Α, δεν σας είχα δει. Ποιετικά είναι. Ευχαριστώ πρώτα. Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ κύριε Υπουργέ διότι νομίζω ότι περιγράψατε πολύ καλά και περιεκτικά τι σημαίνει το πρασίνισμα της οικονομίας. Ότι δεν πρόκειται για αγώνα κατά της βιομηχανίας και υπέρ του περιβάλλοντος, ούτε κατά συγκεκριμένων τομέων της βιομηχανίας. Είναι ένα ζωτικό θέμα που θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, καινούργια έσοδα, ανταγωνιστικότητα και ευημερία για τους Ευρωπαίους. Είναι λοιπόν ένας αγώνας ίσως μεταξύ εταιριών στον ίδιο τομέα. Το καθήκον σας, το δύσκολο καθήκον σας θα ήταν πώς να κάνουμε τη μεταρρύθμιση και τα περιγράψατε πολύ καλά και σαφώς. Resource efficiency. Ε, Επανέρχομαι στο θέμα της ανακυκλούμενης οικονομίας Ίσως να μην κατάλαβα καλά τι είπατε ακριβώς γι' αυτό, αλλά θέλω να θίξω τρία θέματα. Πρώτον, την ενεργειακή αποδοτικότητα. Είστε υπέρ του ορίου του 40%. Και πώς νομίζετε ότι το Συμβούλιο θα τοποθετηθεί επ' αυτού θα συμπεριληφθεί στην οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεύτερον, για την ανακυκλούμενη. Νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε ώστε να υπάρξουν αξιόπιστοι δείκτες για αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ξέρουμε ότι για τη σταθερότητα της αγοράς απαιτούνται τρία χρόνια, αλλά θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε ότι θα εργαστείτε και για το να μην ξαναρχίσουν όλα από την αρχή από το 17. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Uh, Mr. Min Αγαπητέ Υπουργέ, όπως ακούστηκε προηγουμένως, στις θέσεις σας για τη νέα κλιματολογική πολιτική για το 2030, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τον φιλόδοξο στόχο της μείωσης κατά 40% των εκπομπών, 30% αύξησης των εναλλακτικών πηγών και μιας και τέθηκε και το θέμα της μείωσης των εκπομπών στις θαλάσσιες μεταφορές. Αναφερθήκατε επίσης και στην αηφορία των οικονομικών δραστηριοτήτων. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη και το ισχυρό πολιτικό μήνυμα που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζοντας την έλλειψη φιλοδοξίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πώς θα μπορέσει να ε, λάβει υπόψη το Συμβούλιο τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διαφέρουν τόσο πολύ. Για τους πράσινους ο συνάδελφος Τέιλορ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την παρουσίασή του. Σκεφτόμουν τα θέματα ανάπτυξης, ένα είδος ανάπτυξης που είδαμε και δεν θέλουμε να βλέπουμε, είναι η αύξηση στον αριθμό των Ευρωπαίων πολιτών που πεθαίνουν από τη ρήπανση. Βάσει της μελέτης της Κομισιόν, 420.000 άτομα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω των αποτελεσμάτων της ρήπανσης του αέρος, της ατμόσφαιρας. Ελπίζω να έχετε κι εσείς την ίδια αγανάκτηση που νιώθω κι εγώ και να το βρίσκετε κάτι απόλυτα απαράδεκτο. Θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνει η Ιταλική Προεδρία για να εξασφαλίσω ότι θα υπάρξει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα σε σχέση με την ε, μείωση των ε, οροφών των εθνικών εκπομπών και αν θα υποστηρίξετε ένα δεσμευτικό στόχο για το 2025 και τη συμμόρφωση όλων των κρατών μελών σε αυτόν τον υποχρεωτικό στόχο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τέιλορ. Και τώρα για κύριο Νάτζη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για, την, για τις ε, προτεραιότητες Ιταλικής Προεδρίας που παρουσιάσατε και σας υποστηρίζω και σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε για την φιλική προς το περιβάλλον οικονομία. Είναι απαραίτητο επίσης να τονίσουμε και μια μορφή κατανάλωση που να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Και φυσικά οι πολιτικές μας πρέπει να υποστηρίξουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αυτό το έχουμε στο μυαλό μας όταν θέτουμε στόχους για το περιβάλλον. Η κλιματική μας πολιτική και η ενεργειακή μας πολιτική δυστυχώς έχουν δημιουργήσει επενδύσεις οι οποίες δεν ήταν δημιουργές αηφόρου απασχόλησης. Ουσιαστικά οδήγησαν στο κλείσιμο επιχειρήσεων λόγω της πολιτικής για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, ιδίως στις νέες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ανατολική Ευρώπη. Αυτές λοιπόν οι θυσίες δεν έτυχαν αντισταθμίσματος και αποζημίωσης, ε, διότι οι ποσοστώσεις έχουν χάσει την αξία τους. Χωρίς λοιπόν μια συνολική συμφωνία αυτές οι θυσίες θα μείνουν χωρίς να έχουν δημιουργήσει καμία βελτίωση. Ξέρουμε πως η παραγωγική ικανότητα έχει αντικατασταθεί από εισαγόμενα προϊόντα ή έχουν μεταφερθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλες χώρες λόγω της διαρροής άνθρακος μέσα εισαγωγικά. Εάν λοιπόν δεν αλλάξουμε αυτές τις πολιτικές δεν μπορούμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Πιστεύω πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη έμφαση αντί στην εμπορία εκπομπών στο να εξασφαλίσουμε πιο αποτελεσματικά τους φυσικούς μας πόρους με την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και με την ανακύκλωση των δευτερευόντων ε, πρώτων υλών μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσει εργασία που να είναι αηφόρου χαρακτήρα. Και ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Θέλουμε να το προωθήσουμε αυτό για να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή μας ε, ανεξαρτησία ή όχι. Δίνω το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει. Και προηγουμένως όμως κύριε Μούτραν. Ναι, συγγνώμη, άκουγα τη σουηδική μετάφραση και δεν σας ε, κατανόησα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι η παρέμβασή σας ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και χάρηκα πάρα πολύ όταν σας άκουσα να μιλάτε για τις εκπομπές που έχουν να κάνουν με τις θαλάσσιες μεταφορές. Εγώ είμαι σκιώδη εισηγήτρια για το θέμα αυτό, το παρακολουθώ από πολύ κοντά και φυσικά με ενδιαφέρει η δράση τη Ιταλική Προεδρία. Μιλήσατε και για τη διάσκεψη τη Λίμα. Είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ιταλική Προεδρία να μπορέσει να εξασφαλίσει κάποια πρόοδο. Θα ήθελα όμω να μπορέσω να πω στου συμπολίτε μου στη Σουηδία όταν γυρίσω εκεί ότι οι Ιταλοί καταβάλουν πραγματικά προσπάθεια ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται στην αιχμή της λόγχης του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής για να μπορούμε πραγματικά να είμαστε ισχυροί στην επόμενη διάσκεψη της Λίμας. Το ερώτημα είναι λοιπόν πώς θα φροντίσετε οι δεσμευτικοί αυτοί στόχοι που επιθυμούμε όλοι να επιτευχθούν. Ποιο είναι το επίπεδο φιλοδοξίας σας. Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες που θα θεσπίσετε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε από αυτή τη διάσκεψη κορυφή την πιο στεναρή δυνατή θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις ε, ερωτήσεις τους, τις πολύ ενδιαφέρουσες. 7-8 λεπτά κύριε Υπουργέ για να απαντήσετε. Θα προσπαθήσω. Τέσσερις ώρες θα χρειαστώ κανονικά, αλλά δέχομαι την πρόκληση την οποία μου θέτεται. Ένα πράγμα να ξεκινήσω λέγοντας. Είμαι ιδιαίτερο ικανοποιημένος γιατί βρίσκω ότι υπάρχει μια σύγκληση απόψεων πάνω στο κύριο θέμα το οποίο είχα παρουσιάσει στην ομιλία μου. Αυτό το της πολιτιστικής αλλαγής, αυτό το της αλλαγής του βήματος, της αλλαγής ρυθμού και της εξέτασης των προβλημάτων του περιβάλλοντος μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το να βλέπουμε το περιβάλλον όχι σαν πρόβλημα, σαν λύση των προβλημάτων των άλλων τομέων. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι το Συμβούλιο από τη μία, η Προεδρία και το Κοινοβούλιο μπορούν να συνεργαστούν παραγωγικά. Τώρα σε επίπεδο λειτουργικό ε, τι μπορούμε να κάνουμε για να μην μείνουμε σε εκδηλώσεις προθέσεων. Ένα μεγάλο τμήμα των θεμάτων τα οποία ασχοληθήκαμε σήμερα ε, θα έλεγα έχουν άμεση σχέση με τη λεγόμενη πολιτιστική αλλαγή. Όταν μιλάμε για κυκλική οικονομία ή ανακυκλώμενη οικονομία, όταν μιλάμε για αποτελεσματική ή αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, μιλάμε για αλλαγή της δομής της οικονομίας η οποία θα πρέπει να υπηρετεί το περιβάλλον. Εγώ λοιπόν εμένω στην ανάγκη για βελτίωση των οικονομικών δικτών, αλλά σεβόμενο το περιβάλλον, σεβόμενοι οικονομικων δικτων αλλα σεβομενος το περιβάλλον. Σεβόμενοι λοιπόν το περιβάλλον ε, εφαρμόζοντας τις αρχές της λεγόμενης ανακυκλούμενης οικονομίας κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να ελαφρύνουμε και τις κοινωνικές πιέσεις. Τι σημαίνει ανακυκλούμενη οικονομία. Σημαίνει χρήση προϊόντων και χρήση πρώτων υλών που στο τέλος της αρχικής τους χρήσης παράγουν απόβλητα τα οποία είναι χρήσιμα σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες η παραγωγή ενός προϊόντος το οποίο στο τέλος της ζωής του δεν μετατρέπεται σε απόβλητο αλλά παραμένει ανακυκλώσιμο σύνεπώς αναχρησιμοποιούσιμο από τη γραμμική οικονομία στην κυκλική οικονομία. Και αυτό δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Γιατί το λέω αυτό κάποια νέα επαγγέλματα δημιουργούνται γύρω από αυτό. Το eco-design, το οικονομικό σχέδιο, είναι τμήμα του νέου παραγωγικού συστήματος, μας δίνει τη δυνατότητα να προδημιουργήσουμε νέα προϊόντα και προς την κατεύθυνση αυτή επίσης Ε, εγγράφεται και η συμφωνία ε, για το κλίμα και την ενέργεια. Το είπαμε προηγουμένως ότι αν πράγματι θέλουμε να καταλήξουμε σε μια φιλόδοξη συμφωνία θα πρέπει να εμείνουμε στην αποδοτικότητα της ενέργειας, στην σωστή της χρήση. Για τις ανανεώσιμες πηγές εμείς στην Ιταλία έχουμε ένα στόχο ανανεώσιμων ιδιαίτερα υψηλό αυτό μέχρι τώρα έχει δημιουργήσει και πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης και στις δικές σας χώρες άλλωστε. Πρόκειται για μια διαδικασία λοιπόν η οποία έχει ξεκινήσει και την οποία ε, ενισχύουμε ε, συνειδητοποιώντας τις διαφορές τις πολιτιστικές που υπάρχουν. Έχω απαντήσει σε αρκετές ερωτήσεις δεν ήμουν εξαντλητικός ίσως, αλλά εν πάση ελπίζω να είπα περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν για την αναδιάρθρωση του ETS. Το είπαμε προηγουμένως. Το ETS για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι πολλές είναι οι χώρες οι οποίες θέλουν να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Αυτό είναι σημαντικό και θα ληφθεί υπόψη. Για το διεθνές κομμάτι τώρα, Ε, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια της μεταρρύθμισης. Εμείς είμαστε επιφυλακ... προσεκτικοί μάλλον σε σχέση με την χρήση των περιοριστικών διατάξεων. Δεν θέλουμε να αποθαρρύνουμε τους επενδυτές και θέλουμε να συνεχιστούν οι επενδύσεις σε πολλούς τομείς πάντα για το θέμα αυτό των ETS, όπως επίσης και για άλλα ερωτήματα τα οποία φτέθηκαν για το πακέτο κλίμα και ενέργεια, έχω την αίσθηση ότι η σωστή ισορροπία θα πρέπει να αναζητηθεί τους επόμενους μήνες με μια διαπραγμάτευση η οποία θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη. Υπάρχουν στην Ευρώπη, όπως είπα, χώρες περισσότερο φιλόδοξες και άλλες λιγότερο φιλόδοξες. Είναι σαφές λοιπόν, όπως συμβαίνει πολύ συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αναζητήσουμε την ισορροπία. Λέμε στην Ιταλία ότι το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Εγώ θέλω το καλύτερο, αλλά όταν αναζητούμε μια κοινή λύση ανάμεσα σε 28 χώρες θα πρέπει ίσως να αρκεστούμε στο καλό. Λοιπόν, ίσως το τέλος το Συμβούλιο να καταφέρει να βρει μια θέση καλή η οποία να μην είναι βέβαια η καλύτερη δυνατή γιατί υπάρχει αναζήτηση της ισορροπίας των θέσεων 28 χωρών πρέπει η διαδικασία αυτή να κλείσει πριν από την διάσκεψη της Λίμα. Μέχρι τις 16-17, όπως το είπαμε στις 16 και 17 Ιουνίου στο Μιλάνο. Για τις πλαστικές σακούλες είναι ένα θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται ε, δίνεται ειδικό βάρος. Να επαναλάβω εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να προωθήσουμε το θέμα για, τα, για τις πλαστικές σακούλες, γιατί συνειδητοποιούμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, όχι άλλης φύσεως. Οι πλαστικές σακούλες μολύνουν, μολύνουν τις θάλασσες, μολύνουν ε, το κλίμα Πρέπει λοιπόν εμείς να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό κυρίαρχα σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Πρέπει να υπάρξουν βήματα προς τα ευρώς, πρέπει να υπάρξει συμφωνία γύρω από αυτό. Το Κοινοβούλιο θέλει συγκεκριμένους στόχους, ενώ το Συμβούλιο προς το παρόν δεν έχει εκφραστεί γύρω από αυτό. Καλό θα είναι στο τέλος του εξαμήνου να έχουμε μία απόφαση η οποία κάθε, θα επιτρέπει σε κάθε χώρα να δώσει κάποιες ενδείξεις αναδιάταξης της χρήσης της πλαστικής σακούλας και να επιτρέψει στις χώρες οι οποίες το επιθυμούν να μπορέσουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς ρυθμούς για την κατάργησή τους. Για τα απόβλητα τα είπαμε ήδη προηγουμένως. Εμείς θα συνεργαστούμε με ένταση και θα προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε το πώς έχουν σήμερα τα πράγματα και να καταλήξουμε σε μια προχωρημένη πολιτική λύση. Ε, ποιοι είναι οι τρεις βασικοί στόχοι, το top, ε, σύντομα θα σας τα ξαναπώ. Καταρχάς συμφωνία το μήνα Οκτώβριο για το πακέτο κλίμα και ενέργεια 2013. Πρέπει να είναι μια πολύ ε, φιλόδοξη ε, συμφωνία και αυτό είναι η βασική μας προτεραιότητα. Είπα κάτι σημαντικό στην αρχή. Απαιτείται μια νέα οικονομική governance στην Ευρώπη, μια νέα οικονομική διακυβέρνηση που να περιλαμβάνει την περιβαλλοντική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εντόπισα επίσης και κάποια επιπλέον θέματα όπως τα γενετικά τροποποιημένα ή πλαστικές σακούλες και ε, το e-look. Νομίζω ότι με τη βοήθειά σας γύρω από αυτούς τους τομείς θα μπορέσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα προς τα εμπρός. Για τα γενετικά τροποποιημένα. Γνωρίζετε ότι στις 12 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε μία πρόταση εμείς θα πρέπει να εργαστούμε στην πρόταση αυτή, έτσι πριν από το τέλος του χρόνου να έχουμε καταλήξει. E, e Για τις ενδοκρινικές ε, διαταραχές ή τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Εμείς περιμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όταν την έχουμε στη διάθεσή μας θα προχωρήσουμε για την αποτελεσματική χρήση των πόρων και για τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Έχουμε συζητήσει στο Μιλάνο γύρω από αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταστεί ένας πολιτικός στόχος. Αν η πολιτική κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και στη διατύπωση στόχων. Αν τυχόν συμφωνήσουν όλες οι χώρες θα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Πάντως εμείς θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Έχει σημασία να έχουμε μια πρώτη συμφωνία στο Συμβούλιο του μηνός Οκτωβρίου. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, ε, αν δεν απάντησα κάτι, είναι πιο δύσκολο εδώ από ότι να παίρνει κανείς το πτυχίο του το απολυτήριό του. Καταλαβαίνω ότι είναι πολλές φορές οι ερωτήσεις ε, ε, είναι εύκολα διατυπωμένες, αλλά παρόλα αυτά είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς σύντομα. Περνάμε σε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα είμαι σύντομη, διότι το θέμα έχει ήδη συζητηθεί. από έναν άλλο συνάδελφο. Εγώ λοιπόν θα επικεντρωθώ ιδιαίτερα στο θέμα της ανακυκλωμένης οικονομίας και στο θέμα της βιώσιμης διατροφής. Θίξατε λίγο αυτά τα θέματα, αλλά μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω. Ιδιαίτερα για το θέμα των ημερομηνιών που αναφέρονται λήξεις, που αναφέρονται στα τρόφιμα. Ιδίω για τα φρούτα και τα λαχανικά που το σύστημα φαίνεται ότι δεν είναι τέλειο. Δεύτερον, θα υποστηρίζατε μία ενωσιακή δράση συλλογής προϊόντων από τους παραγωγούς που δεν φτάνουν μέχρι τις αγορές ώστε να χαριστούν, να δωρηθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και τρίτον η διαφάνεια των τιμών. Τι θα υποστηρίξετε, τι δράση θα υποστηρίξετε για τις εισαγωγές προϊόντων χαμηλού κόστους, ιδιαίτερα φρουτολαχανικά. Γιατί εδώ τίθεται το πρόβλημα των εσόδων των παραγωγών. Και τι θα τα κάνουν αυτοί τα προϊόντα τους που παραμένουν απούλητα. Λάινεν από τους σοσιαλιστάς. Κύριε Υπουργέ, ήσασταν μέλος της πλατφόρμας, της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων και πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχει μεγάλη κατασπατάληση φυσικών πόρων. Θέλω να σας ε, παροτρύνω να θεσπίσετε ένα συγκεκριμένο στόχο, όπως και στην περίπτωση κλιματικής αλλαγής και για την προστασία των φυσικών πόρων χρειαζόμαστε χρονοδιάγραμματα και συγκεκριμένους στόχους, αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε επιτυχία. Θα ήθελα να ξέρω τι προτείνετε να κάνετε και εν συντομία ένα δεύτερο ερώτημα το Ταμείο για την ε, Κλιματική Αλλαγή, το Πράσινο Ταμείο, είναι ουσιαστικά άδειο. Η Ιταλία θα κάνει κάποια προσπάθεια να συλλέξει νέα κονδύλια για αυτό το Ταμείο. Η Γερμανία υποσχέθηκε 750 εκατομμύρια για αυτό το ταμείο στη συνάντηση του Βερολίνου, παραδείγματος χάρη. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάτεμακή δεν τη βλέπω όμως. Πάω στους πράσινους. Ο Γκάμπορ Σλέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Βλέπουμε ότι Υπάρχει μια συμφωνία σε σχέση με την αντιμετώπιση της ρήπανσης ατμόσφαιρας που είναι φυσικά ένα διαμεθοριακό πρόγραμμα και, πρόβλημα και έχει μεγάλη επίπτωση στο περιβάλλον. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τη χλωρίδα και την πανίδα. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι που στην ε, περιοχή του Σλοβένσκι Μπροντ στην ε, ε, Κροατία είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα με την με, χημικά, με ρήπανση η οποία προερχόταν από την Βοσνία. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας, ρωσικού χαρακτήρα, μιας ρωσικής βιομηχανίας που είχε κατασταθεί εκεί, η οποία δεν είχε εξυγχρονιστεί. Επίσης, συνεχίζει η χρήση του άνθρακα ως καυσίμου και <clears throat> εδώ δεν λαμβάνεται υπόψη η θέση της Κροατίας. Η Βοσνία ζεγοβιν δεν έχουν εγκρίνει μια τέτοια αρρύθμιση για στο κοινοβούλιο του, Θα ήθελα, ξέρω, η Ιταλία σε ποιο βαθμό ως Προεδρία θα μπορούσε να βοηθήσει την Κροατία, μια χώρα μέλος, για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα το οποίο διαιωνίζεται. Ένα πρόβλημα με μια τρίτη χώρα η οποία δεν είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Παολούτσι δεν είναι εδώ. Καπούτο Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Καπούτο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα είμαι σύντομος. Προέρχομαι από την ε, Καμπανία, από την περιοχή με τα Ηφαίστεια, Ξέρετε ότι έχουμε πάνω από 218 παράνομες χωματερές στην περιοχή μου. Και διαρωτώ με τι πρωτοβουλίες θα αναλάβει η Ιταλική Προεδρία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της έτσι ώστε να υπάρξει μια πραγματική στρατηγική αποκατάστασης των περιοχών αυτών που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα με τα σκουπίδια στην περιοχή μας και το οποίο έχει η γνώση και η φήμη του ξεπεράσει τα σύνορα. Οι άλλοι συνάδελφοι δεν είναι παρόντες που είχαν ζητήσει το λόγο και γι' αυτό θα δώσω αμέσως το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει και θα περάσουμε στην επόμενη ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα για την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Το θέμα της πατάλης στον τομέα των τροφίμων συνδέεται με αυτό που είπατε. Μου έχει κάνει εντύπωση γιατί στην Ιταλία ξεκινήσαμε μια έρευνα πάνω στο θέμα αυτό και τα δύο τρίτα των Ιταλών ε, δεν ε, συμπεριλάμβαναν τη σπατάλη των πόρων στα περιβαλλοντικά θέματα. Θεωρούσαν ότι είναι οικονομικό πρόβλημα, ότι είναι κοινωνικό πρόβλημα, αλλά όχι περιβαλλοντικό. Έχουμε λοιπόν μια τεράστια πολιτιστική εδώ πρόκληση, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ότι όταν πετάμε ένα κομμάτι ψωμί, είναι σαν να πετάμε ένα κομμάτι από το περιβάλλον μας, ένα κομμάτι από τους φυσικούς μας πόρους. Εμείς θα, κάνουμε, θα οργανώσουμε μία συνάντηση στις 24 Νοεμβρίου ειδική πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Αξίζει να εμβαθύνουμε και είμαι βέβαιος ότι ένα από τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε για να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο αυτό πρόβλημα είναι να αλλάξουμε την περιβαλλοντική μας αντίληψη, τον περιβαλλοντικό μας πολιτισμό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο από ό,τι ε, μέχρι σήμερα. Γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι ε, θα δημιουργήσουμε περιβαλλοντικά αναλφάβητους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι πάρα πολύ μορφωμένοι σε άλλα θέματα αλλά δεν θα είναι ικανοί να ξεπεράσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ο σεβασμός του περιβάλλοντος είναι βασική αξία λοιπόν για το, την οποία θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε για τα λεγόμενα green food, τα πράσινα τρόφιμα. Εμείς συνεργαζόμαστε με τις υποανάπτυξη χώρες στενά και σε διμερή σχέδια και σε πολυμερή προγράμματα και θα συνεχίσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή όπως πάντα. Για τα γενετικά τροποποιημένα, ίσως δεν έδωσα μια πλήρη απάντηση πριν να συμπληρώσω τώρα. Θέλω να επαναλάβω ότι εμείς από τις επόμενες ημέρες ήδη θα αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε το ταχύτερο δυνατόν σε μια κοινή θέση. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεργαστούμε με, την εισηγήτρια για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση γρήγορα. Για το πρόβλημα της Καμπανίας ε, είναι γνωστό. Εγώ θα πάω στο Καστέλ Βολτούρνο κοντά στην Άπολη ε, μαζί με τον υπεύθυνο Υπουργό είπαμε ότι δεν θέλω να μιλήσω για τοπικά θέματα τώρα. Σας ευχαριστώ πάντως για την υποδοχή σας και τη διάθεσή σας. Ελπίζω να μπορέσω να συνεργαστώ μαζί σας σωστά τους επόμενους έξι μήνες και νομίζω ότι και εμείς και εσείς έχουμε μπροστά μας ότι η δουλειά είναι δύσκολη αλλά οι προσδοκίες υψηλές. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ Γκαλέτη και εμείς κύριε Υπουργέ σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε να σας βομβαρδίσουμε με ερωτήσεις και διακόπτουμε για πέντε λεπτά για να συνοδεύσω τον ένα υπουργό και να υποδεχθώ τον επόμενο. Cari colleghi, colleghi se prendiamo posto Sinadelfi. cominciamo questa seconda audizione. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ακρόαση. Βρες Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ακρόαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό Υγείας της Ιταλίας, την φίλη Μπεατρίτσε Λορεντσίνη, για την παρουσία της ενώπιον της Επιτροπής μας. Μετά από την πρώτη ακρόαση που κάναμε του Υπουργού Γκαλέτη, είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ερωτήσεων που έθεσαν από τους συναδέλφους και θα σας δώσουμε, θα έχουμε την ίδια ε, διαδικασία. Θα σας δώσουμε 10 λεπτά για να εκφράσετε τις βασικές προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας με δύο, και θα ακολουθήσουν δύο γύροι ερωτήσεων. Πρώτα από τους συντονιστές των ομάδων αυτούς που ασχολούνται με το θέμα αυτό μέσα στην ε, πολιτική τους ομάδα και μετά θα υπάρξει ένας δεύτερος γύρος από τους άλλους συναδέλφους μέσα στην Επιτροπή ε, περιβάλλοντος. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για να περάσετε αμέσως στο περιεχόμενο της ε, Ιταλικής Προεδρίας. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος. Σαν υπεύθυνοι για τον τομέα της υγείας που ε, θα κατευθύνουμε αυτό το εξάμεινο της προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας παρουσιάσω το πρόγραμμα το εξαμηνιαίο της Ιταλικής Προεδρίας. Θα μπορέσουμε να κάνουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε αυτούς τους 4,5 μήνες που έχουμε μπροστά μας να θέσουμε τις βάσεις για ένα καινοτόμο πρόγραμμα ε, για τα επόμενα χρόνια συνδυαζόμαστε με τη Λετωνία και το Λουξεμβούργο τους επόμενους 18 μήνες και με τους συναδέλφους των χωρών αυτών προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια των εργασιών του Συμβουλίου και να μην υπάρχουν διακοπές από τη μία χώρα στην άλλη. Στόχος είναι να σχεδιάσουμε μια σωστή πρόταση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασισμένη στην, στην πράσινη οικονομία στα πλαίσια της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Θα αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα τα σημαντικά στον τομέα της πρόληψης του προγραμματισμού για να περάσουμε επίσης και στα θέματα της θεραπείας και της ευημερίας των ζώων. Προσπαθήσαμε εμείς να προχωρήσουμε ε, κληρονομώντας από την Ιταλική Προεδρία ε, και κάποια θέματα τα οποία είναι ακόμα υποσυζήτηση. Η Ιταλική Προεδρία θα συνεχίσει ε, την επικοδομητική της στάση σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο βασικός στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα πιο αποτελεσματικό το οποίο ε, να μας επιτρέψει την περαιτέρω χρήση, ανάπτυξη μάλλον, των ε, ε, τομέων στους οποίους η Ευρώπη είναι leader, είναι ηγέτης. Στις 19 Δεκεμβρίου θα γίνει στη ναι. Ρώμη και η συνάντηση για τους ιατρικούς εξοπλισμούς δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε δύο προτάσεις κανονισμού που είναι υπό εξέταση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς, η αναθεώρηση της οδηγίας για τους ελέγχους που γίνονται λαμβάνοντας υπόψη και για τα τρόφιμα και για τις ζωοτροφές. Ε, και ασχοληθούμε ταυτόχρονα και ό,τι επηρεάζει γενικότερα τον τομέα των τροφίμων και τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, της, οποίους, ε, της οποίας μάλλον αγοράς τους πρωταγωνιστές θα αντιμετωπίσουμε ισότιμα. Αυτά έχουν συζητηθεί και στο παρελθόν και με την ε, προηγούμενη Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Περιβάλλον, την ΕΝΒΗ. Απαιτείται να ξεκινήσουμε το ταχύτερο δυνατόν λοιπόν τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να καταλήξουμε σε, ε, ένα, σε μια δεύτερη ανάγνωση γρήγορα. Η καταπολέμηση των απατών τώρα και υπό το φως των κατευθυντηρίων γραμμών του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την, για την τροφιμική κρίση και τις απάτες στα τρόφιμα που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2013 και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα οργανώσουμε στη Ρώμη μια συνάντηση για τις απάτες στον τομέα των τροφίμων για να αξιολογήσουμε σωστά τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα αυτό. Βασικός στόχος είναι να διατυπώσουμε ένα κοινό προσανατολιστικό κείμενο για το Συμβούλιο. Επίσης σημαντική είναι η πρόταση στον τομέα του novel food, των νέων τροφίμων που θέλει την αναθεώρηση και ενημεροποίηση της οδηγίας και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον εναρμονισμό των διαδικασιών αδειοδότησης κυκλοφορίας προϊόντων. Ο έλεγχος επίσης ε, ε, τον, ε, του σεβασμού των διαδικασιών για το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων είναι κάτι που θα μας απασχολήσει φυσικά. Η διασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας των τροφίμων είναι σημαντική για όλους η Προεδρία εξετάζει αυτή τη στιγμή με θετικό πνεύμα μια κεντρική διαδικασία διοδότησης μετά από αξιολόγηση της ασφάλειας του προϊόντος άμεσα από την ίδια την ΕΦΣΑ. Γνωρίζουμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη στο εσωτερικό του Συμβουλίου. Η Ιταλική Προεδρία θα υπογραμμίσει για μια ακόμη φορά την σημασία που έχουν οι εμβολιασμοί στη στρατηγική της δημόσιας υγείας, θα εξετάσουμε τις νέες προτάσεις για εμβόλια και θα δούμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος των εμβολίων στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε προχωρήσει λοιπόν στην διατύπωση ενός εγγράφου για τα εμβόλια κατά πολλών ασθενειών είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει ε, όχι μόνο αυτούς ε, οι οποίοι ε, έχουν εμβολιαστεί, αλλά στα πλαίσια της γενικότερης δράσης και αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Επίσης θα προχωρήσουμε στην εξέλιξη το, της κατάστασης των πραγμάτων στον τομέα της καταπολέμησης των μολύνσεων ένα τρίτο θέμα το οποίο θα πρέπει να είναι η βάση για μια πρόταση είναι οι θεραπευτικές καινοτομίες υπέρ του ασθενούς. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι περιλαμβάνεται σε αυτήν την έννοια ε, και η καινοτομία στον φαρμακευτικό τομέα, στον τομέα του ιατρικού εξοπλισμού και επίσης ε, η προσωποποίηση κατά κάποιο τρόπο της χορήγησης τροφίμων και η μείωση του κόστους. Ε, σαν παράδειγμα ε, η εφαρμογή των μέτρων αυτών στον τομέα των χρόνιων μορφών υπατήτηδας είναι μια ανησυχία για τις δημόσιες αρχές. Ε, θα ασχοληθούμε επίσης και με τα θέματα αυτά στην ανεπίσημη συνάντηση των Υπουργών στις 22 Δεκεμβρίου. Στις δύο τελευταίες συναντήσεις Υπουργών Υγείας ζητήθηκε μια μεγαλύτερη αντιπροσώπευση και παρουσία της υγείας στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και γι' αυτό ζητάμε ε, μια στενότερη συνεργασία με την Επιτροπή Προστασίας ε, της κοινωνικής, ε, του κοινωνικού τμήματος αν θέλετε που αφορά την υγεία η σχέση ανάμεσα στην οικονομία και την υγεία είναι κάτι το οποίο έχει έρθει στην επιφάνεια σε όλα τα κράτη-μέλη πλέον, όπως επίσης και η ανάγκη να θεωρηθεί η υγεία σαν κάτι το οποίο δεν είναι ένα οριζόντιο κόστος και όχι μια απλή επένδυση για τις κοινωνίες μας. Σχετικά τώρα με την ποιότητα και την επίδοση των συστημάτων υγείας, εμείς ε, θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στον εντοπισμό δικτών που θα χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τις επιδόσεις τους με συγκρίσιμο τρόπο θα ασχοληθούμε και με επιμέρους θέματα όπως η πρόληψη στον τομέα της αποφυγής όγκων, δημιουργίας όγκων μέσω σωστών τρόπων ζωής. Οι καρκινικοί όγκοι μαζί με τις καρδιαγκιακές παθήσεις είναι πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα τρίτο θέμα είναι η αντιμετώπιση του πόνου, η θεραπεία του πόνου και οι τελικές φροντίδες ή η διαδικασία της τελικής φροντίδας. Θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλα θέματα όπως η αντιμετώπιση των προβλημάτων του διαβητικού ασθενούς, η αντιμετώπιση των χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων κτλ. Η πρώτη συνάντηση στις 2 και 3 Οκτωβρίου στη Ρώμη θα έχει σαν στόχο την υγεία των ε, γυναικών ε, με μία αντιμετώπιση μέσω της μεθόδου Life Course. Αυτό είναι κάτι που έχει σχέση σε μια σύγχρονη κοινωνία, ε, την προστασία της υγείας, την αποφυγή παθολογιών, την προστασία της μητρότητας, και επίσης την προστασία των ιδιαίτερα ηλικιωμένων συμπολιτών μας που είναι κυρίως γυναίκες βέβαια. Η συνάντηση αυτή λοιπόν θα είναι μια ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για την υγεία των γυναικών σε όλες τις φάσεις της ζωής τους. Στυλ ζωής, άσκηση, γενετήσια υγεία, αποφυγή ενδομητριώσεων, όπως επίσης και η υγεία πριν, κατά και μετά την γένα. Αντιμετώπιση επίσης των όγκων που επηρεάζουν κυρίως την γυναίκα και ε, προστασία της γονιμότητας σε ασθενείς από όγκους. Νομίζω ότι ένα άλλο θέμα είναι η ψηφιακή υγεία. Εμείς στις 7 και 8 Οκτωβρίου στη Ρώμη ε, θα έχετε την ευκαιρία να έλθετε και να παρακολουθήσετε την σύγκριση των στρατηγικών αυτών ανάμεσα στα κράτη-μέλη στον τομέα της e-health, της ηλεκτρονικής υγείας και των, της παροχής ε, ε, υπηρεσιών μέσω υπολογιστών. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι η προστασία της υγείας στην Μεσόγειο. Η Μεσόγειος είναι μια ευκαιρία για την προώθηση ε, της συνεργασίας για τη δημιουργία μιας υγιούς και ευημερούσας περιοχής. Ε, πρέπει να προχωρήσουμε στην προώθηση λοιπόν των μέτρων που θα διασφαλίσουν την υγεία των πληθυσμών της περιοχής. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες χώρες και είναι θα έλεγα και μια ευκαιρία οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που θα ευνοήσει την επιστροφή της ειρήνης και θα βοηθήσει να ξεπεραστούν τα πολιτιστικά και οικονομικά προβλήματα. Στις 3 Νοεμβρίου θα γίνει και η διάσκεψη ε, για την ποιότητα και το κόστος των θεραπείων. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό για την Προεδρία μας και θα, κάνουμε, θα ξεκινήσουμε πολλές πρωτοβουλίες γύρω από αυτό. Θα συνδέσουμε ε, την αποδοτικότητα την κλινική και την οργανωτική με την αποδοτικότητα την οικονομική. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό για όλα τα συστήματα υγείας για να συνδυάσουμε την δυνατότητα της, της συντήρησης των συστημάτων αυτών και της ποιότητας των, των μεθόδων θεραπείας για την άνοια επίσης θα ε, κάνουμε μια συνάντηση η οποία λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής είναι ένα όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συζητήσουμε τα θέματα τα οποία συνδέονται με τις διάφορες εκφάνσεις της άνοιας και θα προωθήσουμε το θέμα γενικότερα της υγείας των ηλικιωμένων. Θα δώσουμε μεγάλη προσοχή και στην διάσκεψη για την καταπολέμηση του AIDS μετά από το Δουβλίνο μετά από 10 χρόνια. Θα ξεκινήσει ε, με την ημέρα την παγκόσμια για την καταπολέμηση του AIDS. Έχουμε σημειώσει σημαντικά βήματα νικηφόρα το τελευταίο καιρό που έχουμε φτάσει στο βιώσιμο, στο προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών από HIV που να είναι ανάλογο με το αντίστοιχο προσδόκιμο των υπολείπων μη ασθενών. Ε, θέλουμε όλα αυτά τα θέματα να τα συζητήσουμε προσεκτικά ε, και με την κοινωνία των πολιτών η οποία εκπροσωπείται σωστά στον συγκεκριμένο τομέα. Δέκα χρόνια μετά από τη διάσκεψη του Δουβλίνου θα πρέπει να δώσουμε μια νέα όφηση για την καταπολέμηση αυτής της ασθένειας. Στις 4 και 5 ε, Δεκεμβρίου θα κάνουμε και μία διάσκεψη ειδική για τα επαγγέλματα της υγείας, για την κατάρτιση των επαγγελματιών στον τομέα αυτό και για τη σωστή του συνεργασία. Στη Βελετία 16 με 18 Δεκεμβρίου θα λάβει χώρα μία συνδιάσκεψη για την η ψυχική υγεία των νέων. Οι νέοι μεταξύ 10 και 24 ετών, όπως ξέρετε, είναι 27% του παγκόσμιου πληθυσμού και πάνω από 27, 75% των ψυχικά διαταραχών εμφανίζονται μέχρι τα 25 έτη ηλικία. Λαμβάνοντα υπόψη ότι εμφανίζονται σε διάφορε φάσει τη ε, ε, εξέλιξη και μέχρι την ηλικία που ενηλικιώνονται, είναι απαραίτητο να υπάρξουν κατάλληλε υπηρεσίε για τα παιδιά και του εφήβου, ώστε να εξασφαλίσουμε την συνέχεια στην θεραπεία του. Ένα άλλο θέμα μεγάλη σημασία σε αυτή την περίπτωση είναι η αντίσταση κατά των ε, μικροβιακών, αντιμικροβιακών και αντιβιωτικών. Προβλέπεται λοιπόν να γίνει μια συνδιάσκεψη για το θέμα αυτό. Αυτή η προβληματική θα αντιμετωπιστεί με την προοπτική του να υπάρχει η λεγόμενη One Health, μία μονάχα αντιμετώπιση για την υγεία που να λάβει υπόψη τα θέματα και της ανθρώπινης και της ζωικής υγείας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην οδηγία 2012-2024 για μια βελτίωση της, της διεθνούς υγείας και θα υπάρξει στις 15-18 Δεκεμβρίου μια συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Θέλω λοιπόν να τονίσω εν κατακλείδη το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο συνομοθέτη για να θεσπίσει τις πολιτικές και στρατηγικές αλλαγές οι οποίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση των πάνω από 500 εκατομμυρίων καταναλωτών και πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική. Μια πολύ σημαντική πρόκληση για όλους μας και έχουμε ενώπιον μας ένα νέο κοινοβούλιο σχεδόν πλήρως ανανεωμένο που αντιμετωπίζει μια νέα εποχή και νομίζω ότι από κοινού μπορούμε να χαράξουμε κοινέ στρατηγικές στον τομέα της υγείας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Θέλω λοιπόν πάρα πολύ να έχω μια σχέση συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Επιτροπή Ένβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να κάνουμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα και χρήσιμα για την υγεία όλων των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Και τώρα... τώρα... Ξεκινάμε λοιπόν με τους συντονιστές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Πέτερλε πρώτος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Συγχαρητήρια. Είπατε πολλά στα 10 λεπτά που διαθέτατε. Σας καλωσορίζω εδώ για δεύτερη φορά ως Υπουργό Υγείας και χαίρομαι που η Ιταλική Προεδρία προμοθεί την υγεία και την πρόληψη και τον υγιή τρόπο ζωής. Ελπίζω η Τρόικα των Προεδριών να ακολουθήσει την αρχή της συνεχείας γιατί κάθε Υπουργός Υγείας πρέπει να έχει στο Υπουργείο του μία υπηρεσία για την υγιεινή ζωή. Οι πολίτες ανησυχούν γιατί ο διαβήτης και οι καρκίνοι αυξάνονται. Αυτό σημαίνει ότι η προληπτική αντιμετώπιση πρέπει να δυναμωθεί. Η προώθηση της υγείας πάντα συμπεριλαμβάνεται στα δικά μας ψηφίσματα και λευκές βίβλους. Αλλά και ο αριθμός των ασθενών αυξάνεται. Ρωτώ λοιπόν, τι χρειάζεται κατ' για να συν τη διακυβερνητική μέθοδο με την κοινοτική και να καταλήξουμε σε κάτι πιο αποτελεσματικό ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να νιώσουν το αποτέλεσμα. Τι θα μπορούσε να προσθέσει αξία σε ενωσιακό επίπεδο γιατί συχνά ακούμε ότι η υγεία είναι δικαιοδοσία των κρατών μελών και έτσι δεν γίνεται τίποτα. Είμαι βέβαιος ότι αν δεν αλλάξει η συνθήκη ε, ότι χωρίς να αλλάξει η συνθήκη μπορούμε να κάνουμε κάτι για την υγεία και ενωσιακός. Χρειαζόμαστε κάποιον που να υψώσει τη φωνή του και να μιλήσει για την πρόληψη στην Κομισιόν ας πούμε. Εσείς θα υποστηρίζατε μια δέσμευση για να αυξηθεί το μερίδιο από το 3 στο 5% της προληπτικής αντιμετώπισης. Κυρία Υπουργέ ο κύριος Γκαλέτη, ο συνάδελφός σας, μας είπε το πρωί ότι τα περιβαλλοντικά πρέπει να συμπεριληφθούν στην, στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, αλλά εγώ νομίζω θα έπρεπε να συμπεριλάβουν και τα θέματα της υγείας. Είναι και αυτό σημαντικός τομέας. Έστειλα ήδη μήνυμα στον, κύριο Γιούνκερ περί αυτού. Τώρα για τους σοσιαλιστές ο κύριος Κουότα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Έχετε αναφέρει πάρα πολλές συνδιασκέψεις, πάρα πολλές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση διαφορετικών ασθενειών και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει και μία συνδιάσκεψη για την άνοια. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κατά πόσο υπάρχει μια στρατηγική για αυτήν την ε, ασθένεια που είναι πιο συχνή όλο και περισσότερο γιατί αυξάνει η μέση ηλικία του πληθυσμού. Αν θα υπάρξει λοιπόν η μια στατική που θα εξέλθει από αυτήν την ε, ε, συνδιάσκεψη για τις ιατρικές συσκευές. Περιμένουμε ακόμα τη θέση του Συμβουλίου. Περιμένουμε να υπάρξει μια θέση για να προχωρήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Ίσως μπορείτε να μας αναφέρετε κάτι για το θέμα αυτό, επίσης και για την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Ο αριθμός των ε, <clears throat> νέων μολύνσεων από μικρόβια στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι αυξάνεται συνέχεια. Τι θα κάνετε σε σχέση με το θέμα αυτό τους 4,5 ουσιαστικά μήνες της Προεδρίας σας. Και τελευταίο, αλλά όχι ίστατο, η TTIP, η συμφωνία TTIP με τις ΗΠΑ Σε ποιο βαθμό θα προσπαθήσετε να εξασφαλίσετε την διατήρηση των προτύπων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση. Ποια είναι η στρατηγική σας για το θέμα αυτό και σε ποιο βαθμό θα εξασφαλίσετε επίσης να εξασφαλίσετε την ε, ε, διατήρηση των συστημάτων αδειοδότησης στην Ευρώπη για μετά από την TTIP, γιατί υπάρχει μεγάλος φόβος στην Ευρώπη ότι θα μειωθούν τα δικά μας πρότυπα και θα εγκριθούν πιο χαλαρά πρότυπα με τη συμφωνία αυτή. Έχουμε πολύ καλά πρότυπα για την αδειοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατανοείται ότι δεν θέλουμε να χαλαρώσουν ή να εισαχθούν νέα πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποιο βαθμό αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αντιμετωπιστεί ή θα αντιμετωπιστεί κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας από τους Υπουργούς Υγείας. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέρλινγκ από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ και εγώ συνεχίζω λιγάκι από εκεί που αναφέρθηκε ο προπροηγούμενος ομιλητής. Μίλησε, ο κύριος Πέτρελε μίλησε για ασθένειες όπως ο καρκίνος. Εγώ αυτό θα αντιμετωπιστει κατα τη διαρκεια της ιταλικης προεδριας απο τους υπουργους υγειας ευχαριστω η κυρια γκερλινγκ απο την ομαδα των συντηρητικων και μεταρρυθμιστων ευχαριστω και εγω συνεχιζω λιγακι απο εκει που αναφερθηκε ο προπροηγουμενος ομιλητης μιλησε ο κυριος Πέτελε μιλησε για ασθενειες οπως ο καρκινος εγω αυτο θα ηθελα να σταθώ σε θέματα πρόληψης και φυσικά για την εξασφάλιση της γενικής υγείας των ε, πολιτών μας και για τις ε, λεγόμενες, τους λεγόμενους ισχυρισμούς ότι ένα προϊόν είναι υγιεινό. Αν έχουμε μια σωστή αξιολόγηση για τις ουσίες αυτές οι οποίες κυκλοφορούν, αν έχουμε την σωστή προστασία των καταναλωτών από απατηλές διαφημίσεις και η γενική θέση είναι ότι δεν το έχουμε πετύχει αυτό ακόμα. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Ιταλούς. Έχω συνεργαστεί με πολλούς Ιταλούς συναδελφούς στο παρελθόν και το γνωρίζω και ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες στον τομέα αυτό. Αυτό το οποίο θα σας ρωτήσω είναι το εξή. Ξέρουμε όλοι ότι θεωρητικά, αλλά βέβαια πρέπει να το επικυρώσει η νέα Κομισιόν, θα γίνει μια αναθεώρηση του κανονισμού για, τις, για τους ισχυρισμούς σε σχέση με την επίδραση στην υγεία των προϊόντων. Θα ήθελα να ξέρω αν η Προεδρία έχει κάποια σχέδια για αυτό το θέμα, κάποια μορφή δημόσιας ε, ε συνδιάσκεψης ή κάποιας ε, τύπου δημοσίων σχέσεων για το θέμα αυτό, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε τους συμπολίτες και καταναλωτές για το θέμα αυτό. Η κυρία Ρίση για την ομάδα των φιλελευθέρων. Σε ευχαριστώ και εσάς κυρία Υπουργέ για αυτή την πλήρη παρουσίαση. Θα επανέλθω σε δύο θέματα που είχα θέσει και στον συνάδελφό σας Καλέτη, αλλά ο οποίος ξέχασε τη μία και παρέλειψε την άλλη. Αυτό που θεωρώ σημαντικό για τους πολίτες είναι η κατασπατάληση των τροφίμων Ξέρουμε πόσες χιλιάδες τόνοι σπαταλούνται κάθε χρόνο στην Ένωση. Δεν θεωρείτε ότι τροποποιώντας κάποια νομοθεσία, ας πούμε για τη σήμανση ή σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές για την ημερομηνία λήξης των τροφίμων, θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε και σε αυτό το αίτημα των πολιτών που είναι πολύ επίγον και τους ενδιαφέρει πολύ. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε αλλά στο πω και εγώ, το είπατε κι εσείς, στο πρόγραμμά σας έχετε τις εκφυλιστικές ε, ασθένειες όπως Αλτσχάιμερ και άλλες ε, ήταν, προεδρία, ήταν προτεραιότητα και της Γαλλικής Προεδρίας και αν δεν απατώμε το 2013 επεξεργάστηκε το πρόγραμμα Αλκόβ ιδιαίτερα για τη συνεργασία με τους συλλόγους και τις οργανώσεις των πολιτών. Είπε δε και ο κύριος Γκρότε ότι χρειάζεται μια ολόκληρη στρατηγική, ένα καινούργιο πρόγραμμα, όχι μόνο διάλογο. Και εκείνοι και εμείς το χρειαζόμαστε. Και καταλήγω λέγοντας ότι η παχυσαρκία δεν εμφαίνεται πια στο πρόγραμμα των προεδριών ενώ είναι από τα, τις μεγάλες πληγές της κοινωνίας μας και δημιουργεί πολλές παθολογίες. 5 με 10% όλων των προϋπολογισμών υγεία όλων των κρατών μελών αφορούν την παχυσαρκία. Πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν αυτό το επίγον πρόβλημα της παχυσαρκίας που δεν είναι καθόλου δευτερεύουν και αφορά και τους νέους. Ας το δούμε η κυρία Φορέντσα για την ΚΟΕ. Καλημέρα κυρία Υπουργέ. Να θέσω ορισμένε ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά ένα θέμα το οποίο ήδη έχει τεθεί από προηγούμενους ομιλητές είναι η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Σαν κοινευτική ομάδα έχουμε ήδη εκδηλώσει την αντίθεσή μας και τις βαθύτατες ανησυχίες μας σχετικά με τους όρους της συγκεκριμένη διαπραγμάτευσης. Θεωρώ ότι η Ιταλική κυβέρνηση θα πρέπει να ε, εκφράσει τις ανησυχίες της γύρω από το θέμα αυτό ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων και συγκεκριμένα στον τομέα των τροφίμων. Πρόσφατα σαν Ιταλίδα άκουσα τον Υφυπουργό Ρότσι να μιλάει για τη συμφωνία αυτή λέγοντας ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ιταλία. Αντίθετα πιστεύω ότι όπως έλεγα και γενετικά τροποποιημένα προηγουμένως η κίνδυνη για τη χώρα μου είναι πάρα πολύ υψηλή. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας ε, σαν Ιταλίδα Υπουργού. Το δεύτερο θέμα αφορά την υγεία των γυναικών, ένα θέμα το οποίο ε, θέσατε ήδη. Νομίζω ότι από το πρόγραμμα του εξαμήνου σας ελείπει η εγγύηση ενός δικαιώματος το οποίο στην Ιταλία βρίσκεται υπό επίθεση και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η εθελοντική δηλαδή διακοπή κοίησης. Ξέρετε ότι πολλές φορές τα Ιταλικά νοσοκομεία ελέγχουν την επιθυμία των γυναικών και θα ήθελα σαν υπουργό να μας πείτε τι μπορείτε να κάνετε γύρω από τον τομέα αυτό. Η τελευταία ερώτηση αφορά την δυνατότητα παρέμβασης στον τομέα της υγείας στο χώρο εργασίας για άνδρες και γυναίκες. Ξέρετε ότι εμείς ε, ε, το δικαίωμα στην εργασία και το δικαίωμα στην υγεία πολλές φορές ε, δεν συνδυάζονται και εδώ αναφέρομαι στη μονάδα Ήλβα στον Τάραντα. Νομίζω λοιπόν τι, ότι πρέπει να μας πείτε τι μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε να διασφαλίσετε την συμβατότητα αυτών των ε, δύο δραστηριοτήτων. Ευχαριστώ η κυρία Άουκεν για τους πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Εμείς προσβλέπουμε σε μια δεσμευμένη και στρατευμένη Ιταλική Προεδρία. Εδώ είμαι. Με ισχυρή στα θέματα υγείας και ένα περιβάλλον χωρίς τοξίνες. Θέτω το ίδιο ερώτημα το οποίο θέσε και ο κύριος Κρότη για, τους, για τις ιατρικές συσκευές, των ιατρικό εξοπλισμό, όπου περιμένουμε δύο πράγματα μας ενδιαφέρουν. Θέλουμε μια διαδικασία έγκρισης φυσικά πριν από την εμπορία, αλλά θα ήθελα να δω αν μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμασιών θα δημοσιεύονται, θα γίνονται διαθέσιμα. Ξέρουμε από τις κλινικές δοκιμές για τα φαρμακευτικά σκευάσματα ότι αν έχουμε πλήρη διαφάνεια και αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι είναι πραγματικά ασφαλείς αυτές οι δοκιμές και αξιόπιστες, αυτό είναι σημαντικό και θέλω, θέλω το συνδέσω και με την συμφωνία TTIP. Ένα από τα βασικά θέματα που θέλαν να εμποδίσουν οι αμερικανικές φαρμακευτικές εταιρείες πριν από τις εκλογές ήταν ακριβώς αυτή η οδηγία για τις κλινικές δοκιμάσεις. και ελπίζω ότι θα έχουμε ένα ισχυρό υπερασπιστή αυτών των θεμάτων σε εσά. Κάτι ακόμα το οποίο συνδέεται με τις με τις ε, ιατρικές συσκευές είναι ότι αυτές οι συσκευές έρχονται σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα και γι' αυτό δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τοξικές ουσίες. Εκτός αν δεν υπάρχει κανένα, καμιά εναλλακτική δυνατότητα και εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε τον καρκινογόνο χαρακτήρα τους, τον μεταλλαξιογόνο, τον τοξικό χαρακτήρα που έχει επιρροή στην αναπαραγωγή. Θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εστίαση μέχρι στιγμή. Ξέρουμε πόσο επικίνδυνα είναι αυτά για την ανθρώπινη υγεία και γι' αυτό το ερώτημα μας είναι μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι και αυτές οι τοξικές μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες ουσίες θα τύχουν όχι μονάχα έρευνας αλλά και θα υπάρξει η δυνατότητα να εμποδιστεί η χρήση του σε ηλεκτρικές συσκευές. Ευχαριστώ πολύ για την FDD ο κ. Πετιτσίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, όπως και πριν για τον Υπουργό Γκαλέτη, σας προτείνω το ίδιο που πρότεινα πριν. Ε, θέσω μία ερώτηση όχι προσωπική. Μια ερώτηση η οποία διατυπώνεται από τους Ιταλούς πολίτες τους οποίους εκπροσωπώ εδώ. Πρόκειται για μια δράση άμεσης δημοκρατίας. Ε, θα φανεί το ερώτημα αυτό σαν κάτι το τοπικό, τοπικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι όμως έτσι. Εγώ κατανοώ ότι γνωρίζετε ότι προερχόμαι από την Καμπανία, πήγα σε μια περιοχή όπου παράγεται ε, πετρέλαιο εργάζομαι στον τομέα της καταπολέμησης των όγκων, καταλαβαίνω τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και αυτό δεν θα πρέπει να δημιουργήσει ένα προηγούμενο και για τις υπόλοιπες χώρες μέλη. Το ερώτημα είναι το εξής λοιπόν, λόγω της κρίσιμης κατάστασης της περιβαλλοντικής ε, όπως ε, στην περιοχή Ήβα, στον Τάραντα, στην Καμπανία, στην Μπαζιλικάτα, στο Σούτσι, στην Σαρδινία και στο Κάπαρο, στην Μπρέσα που συνδυάζουν ε, προβλήματα περιβαλλοντικά πολλαπλών τύπων όπως και παράνομες χωματερές τοξικών υλικών Όλα αυτά δείχνουν ότι η Ιταλία δεν είναι ικανή να προστατεύσει το επίπεδο των υδάτων που προορίζονται για χρήση από τους ανθρώπους, ιδιαίτερα στην περιεκτικότητα σε φθόριο και σε ε, ε άλλες χημικές επικίνδυνες ουσίες όπως το ασθενικό. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω πως αυτό το οποίο εσείς ε, παρουσιάσατε, ότι δηλαδή πρέπει να προωθήσετε ε, στυλ ζωής ε, καλύτερα για την υγεία, δεν σημαίνει τίποτα γιατί υπάρχουν προβλήματα περιβαλλοντικά που προκαλούν όγκους, φυσικά στον τομέα αυτό, και το θέμα δεν είναι ιταλικό, δεν είναι εθνικό, πρέπει να δούμε αν πρέπει να δημιουργήσουμε μητρώα όγκων. Ε, δυστυχώς τα δεδομένα που συλλέγονται στην χώρα μου είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η Ιταλική Προεδρία για να μπορέσει να θέσει σε εφαρμογή την Ευρωπαϊκή Αρχή που λέγει ότι όποιος μολύνει πληρώνει. Ευχαριστώ λοιπόν τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις τους. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Υπουργό Λορεντσίνα η οποία έχει συμπληρώσει πάρα πολλές σελίδες απαντήσεων, δεν ξέρω αν στο χρόνο που έχει, στα 6-7 λεπτά, θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις. Για την πρόληψη. Είναι ένα θέμα το οποίο καλύπτει θα έλεγα πολλές άλλες ερωτήσεις. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι η πρόληψη είναι το στρατηγικό όπλο υπαριθμένα για την καταπολέμηση των μη μεταδοτικών χρόνιων ασθενειών και εναντίον φυσικά των μεταδοτικών ασθενειών το να ε, επενδύει κανείς στην πρόληψη είναι μια προτεραιότητα σημαντική για όλους. Εμείς επενδύουμε αυτή τη στιγμή ε, το 3% των μέσων μας ε, στην πρόληψη. Είναι ένα χαμηλό ποσοστό σε σχέση με τις ανάγκες που έχουμε. Όλες οι επιστημονικές μελέτες και όλες οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες δείχνουν ότι το μεγαλύτερο τμήμα των μη μεταδοτικών χρόνιων ασθενειών οφείλονται σε, μια κακή, ε, σε ένα κακό τρόπο ζωής. Διατροφή, ε, κάπνισμα, αλκοόλ, ε, ουσίες, ε, έλλειψη γυμναστικής και αθλητισμού. Ξέρουμε ότι ε, το να έχει κανείς ένα σωστό τρόπο ζωής παίζει σημαντικότατο ρόλο στον διαβήτη σαν παράδειγμα που οφείλεται στα τρόφιμα. 30 λεπτά άσκηση την ημέρα βελτιώνουν πάρα πολύ την κατάσταση. Ένα σωστός τρόπος ζωής για ένα ασθενή που έχει διαβήτη ε, σημαίνει ότι θα εξοικονομήσουμε τρία δις σε φαρμακευτική δαπάνη. Μιλάμε δηλαδή και για πολύ σημαντικούς αριθμούς αν τους συγκρίνουμε με το ευρύτερο πλαίσιο. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι απαιτείται μια σωστή στρατηγική για το σύνολο της Ένωσης. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την πρωτοβάθμια πρόληψη ε, και για την ε, ε, δεύτερη φάση βέβαια με τα screening, τους ελέγχους κτλ. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε εμείς ακριβώς την ζωή μας είναι οριζόντιες ορισμένες πολιτικές και είναι μια καλή απάντηση στο πρόβλημα της αηφορίας των συστημάτων υγείας μας. Από τη μία έχουμε λοιπόν την ανάγκη να κάνουμε τα συστήματά μας αποδοτικά, να αντακαταστήσουμε ανταγωνιστικά παρά τη μείωση των πόρων την οποία όλοι γνωρίζουμε και συναντάμε τα τελευταία χρόνια και ταυτόχρονα πρέπει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητά τους. Δεν θα είναι επαρκές να ισορροπήσουμε εμείς το ύψος των διαθεσίμων πόρων με τις ανάγκες μας. Πρέπει να προωθήσουμε νέα προγράμματα πρόληψης. Η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολλά γι' αυτό. Συζητώ, μιλώντας με μία φωνή, με ενιαίο τρόπο, καθιστώντας το, την ιδέα του να φροντίζει κανείς τον εαυτό του κάτι το, ε, το πολιτιστικό, κάτι το κοινωνικό. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα πάνω στο οποίο πρέπει ε, να επενδύσουμε. Το να περάσουμε από το 3 σε 5% του προϋπολογισμού είναι ένα τεράστιο βήμα και θα πρέπει να δούμε πώς θα το πετύχουμε. Γι' αυτό λοιπόν και απαντώ εδώ σε μια άλλη ερώτηση και δεν θυμάμαι ποια είναι, είναι η σχέση με την οικονομία. Όχι μόνο το θέμα του περιβάλλοντος είναι κάτι το οποίο διαπερνά το σύνολο των οικονομιών και της οικονομίας της υγείας. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχουν διαφορές και είναι σωστό που η Επιτροπή σας αφορά το περιβάλλον και την υγεία, γιατί η υγεία είναι η ευημερία. Εμείς μιλάμε για νέα συστήματα υγείας σήμερα. Ε, δεν μιλάμε για την απουσία μόνο της ασθένειας, αλλά κάτι περισσότερο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο λοιπόν τα δύο θέματα αυτά, η υγεία των ανθρώπων, η υγεία των ζώων, οι τροφές μας, οι ζωοτροφές, ο αέρας, το νερό και ο σεβασμός του περιβάλλοντος στο οποίο κινούμεθα. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε έτσι ώστε να είναι ε, συμβατές οι ε, ενέργειές μας με τους στόχους που έχουμε για την επιβίωσή μας. Και εδώ θα μας βοηθήσουν και οι νέες τεχνολογίες. Έχει υπάρξει ένα τεχνολογικό άλμα στον τομέα της υγείας, στον τομέα της πρόληψης και αυτό είναι καθοριστικό για το τι μπορούμε να κάνουμε στην συνέχεια. Παραμένω στο προηγουμένο στο θέμα της ανθρώπινης υγείας, ε, το οποίο έχει ήδη Το θέμα σαν παράδειγμα soprattutto dell'obesità infantile. Της παχυσαρκίας. Ε, δεν είναι απλά ένα πρόβλημα, είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που, που εξαπολύουν διάφορες ασθένειες λόγω της κακής ε, πρόληψης. Η καλή πρόληψη σημαίνει ότι προλαμβάνουμε την παχυσαρκία των παιδιών. Το βλέπουμε αυτό σήμερα ότι υπάρχει κατά τη διάρκεια της κοίησης η κατάλληλη ε, εκπαίδευση των μελλοντικών μητέρων για τον τρόπο με τον οποίο η δική τους διατροφή θα έχει επιπτώσει στη διατροφή του βρέφους τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επιπλέον, όπως δείχνουν οι νέες μελέτες, το είδος ε, ζωής που περνάει ένα παιδί τους πρώτους χρόνους της ζωής του και που επηρεάζουν και τη συνέχεια των διατροφικών του συνήθειών. Η πολιτική λοιπόν που πρέπει να συζητήσουμε και όχι μοναχά στις που είναι πολύ ευχάριστο να έρθετε και στην πόλη μου στη Ρώμη και όχι μόνο στο Μιλάνο για να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να τα εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε και το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι το θέμα των διαφόρων μορφή άνοια. Υπήρξε ένα σχέδιο κατά τη διάρκεια τη γαλλική προεδρία και επίσης τον Δεκέμβριο στο Λονδίνο θα συζητήσουμε για μια γενική στρατηγική για τις διάφορες μορφές άνοιες, είναι απαραίτητο να έχουμε και μια σωστή κατεύθυνση και, μια, και ένα σχέδιο δράσης και πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε νέα στοιχεία που θα προέλθουν από τις ε, από την επιστήμη για τις ασθένειες αυτές όπως είναι το Alzheimer που είναι μια μάστιγα για όλους μας τα επόμενα χρόνια αλλά συγχρόνως εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες να ξεκινήσουν αυτά τα ε, προγράμματα τα οποία θα έχουν επιρροή στη δημόσια υγεία. Το θέμα της TTP της ε, συμφωνίας υποδιαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η διαπραγμάτευση είναι κάτι το οποίο ε, με έχει απασχολήσει και εμένα ως Ιταλίδα Υπουργό στη Νέα Υόρκη. Η διαπραγμάτευση πρέπει να γίνει επί τη βάση επιστημονικών πορισμάτων και αυτό λέγεται και στο σχέδιο συμφωνίας ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ποιοτικά στοιχεία από τις κλινικές δοκιμασίες και στην Ευρώπη μας ενδιαφέρει να έχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας και θα δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή σημασία στο να εξασφαλίσουμε ότι η υγεία των πολιτών μας θα είναι ένα παράγραπτο και μη υποκείμενο σε διαπραγμάτευση στοιχείο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν στερεές επιστημονικές βάσεις για οτιδήποτε συμφωνηθεί και αυτά θα είναι στοιχεία που θα αντιμετωπιστούν και από την ΕΦΣΑ και άλλους φορείς. Είναι μια ευκαιρία η TTTP και νομίζω ότι η Ευρώπη έχει το ειδικό βάρος για να μπορέσει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και ένα ρόλο ίσου για την διαπραγμάτευση αυτή σχετικά με τις πατάλες στον τομέα των τροφίμων. Είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Εγώ προσωπικά το έχω αντιμετωπίσει και σαν βουλευτής στην Ιταλική Βουλή γιατί στην παρούσα φάση η σπατάλη των τροφίμων είναι κάτι το οποίο δεοντολογικά είναι απαράδεκτο. Όταν σκεφτεί κανείς το πόσο έχει αυξηθεί η φτώχεια στους πληθυσμούς μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την αναθεώρηση του κανονισμού 178 του 2002 για να επιτραπεί η χρήση τροφίμων που διατηρούν ορισμένα χαρακτηριστικά υγείας, υγιεινής, αν και για εμπορικούς λόγους ε, ε, φεύγουν από την αγορά των προϊόντων η πρόταση που κάνουμε για την επεξεργασία και την δυνατότητα χρήσης προϊόντων πέρα από την ημερομηνία λήξης είναι μια σκέψη η οποία μας απασχολεί. Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις σας, απαντώ πολύ συνοπτικά. Ας πάμε τώρα στους ιατρικούς εξοπλισμούς. Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω ορισμένα θέματα όπως σαν παράδειγμα η αντίσταση στα μικρόβια Εδωτίθεται το θέμα της σωστής χρήσης των φαρμάκων και της πρόληψης. Το Δεκέμβριο στη Ρώμη έγινε μια συνάντηση του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας για την αντίσταση στα αντιμικροβιακά φάρμακα και αντιβιωτικά. Η ανθρώπινη, το, το σώμα έχει αρχίσει να μην ανταποκρίνεται στις θεραπείες, κάτι το οποίο θίγει φυσικά την υγεία των προσώπων. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα προγράμματα δράσης, χρησιμοποιώντας με σωστό τρόπο τα αντιβιωτικά και να χρησιμοποιήσουμε νέες καινοτόμες τεχνολογίες στα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση των νέων ιών και να δώσουμε επίσης κίνητρα και στην καινοτομία στον τομέα των αντιβιωτικών. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε δράση και σε σχέση με τους ασθενείς και τους, ε, επίσης και, τα, και στον τομέα των κτηνιατρικό. Έχουμε ανάγκη από κατευθυντήριες γραμμές εθνικές αλλά και διεθνείς που θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε μια διαδικασία σημαντικότατη για την ασφάλεια των ασθενών ε, και φυσικά και για την υγεία στον τομέα των τροφίμων. Τώρα για τους ιατρικούς εξοπλισμούς. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο και σημαντικό. Είναι ένα θέμα στο οποίο συναντάμε θέσεις οι οποίες μεταξύ τους δεν είναι συμβατές. Το ισχύον νομικό πλαίσιο έχει δείξει ότι έχει θετικά στοιχεία, αλλά έχει υποστεί και κριτική. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ιατρικό υλικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολόγησε τις προτάσεις οι οποίες είχαν γίνει και στην πρώτη ανάγνωση στο, προς το Συμβούλιο, με το Συμβούλιο έγιναν 35 συναντήσεις της ομάδας εργασίας ε, κάτω από την Λιθουανική, την Κυπριακή και την ελληνική προεδρία. Απαιτείται λοιπόν να αναλυφθεί δράση έτσι ώστε να ενισχύσουμε τον έλεγχο γύρω από την κυκλοφορία αυτών των ιατρικών εξοπλισμών. Η Ιταλική Προεδρία προγραμματίζει μια ε, έντονη δραστηριότητα του Συμβουλίου σε επίπεδο τεχνικών ομάδων. Έχουμε στείλει ερωτηματολόγια σε όλες τις χώρες και τώρα έχουν αρχίσει να επιστρέφονται κάποιες απαντήσεις. Ε, βασικός μας στόχος είναι να προσπαθήσουμε να ορίσουμε μέχρι το τέλος του φθινοπόρου ένα κείμενο που θα γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των κρατών μελών και θα αντιπροσωπεύει τις θέσεις του Συμβουλίου. Τέλος, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υγείας στις 20 Ιουνίου, οι περισσότεροι από τους Υπουργούς Υγείας των κρατών μελών εξέφρασαν την ευχή να κλείσει το θέμα κατά τη διάρκεια της δικής μας Προεδρίας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν από κοινού να εργαστούμε, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια συμβιβαστική λύση έτσι ώστε να δώσουμε εγγυήσεις για ένα κείμενο το οποίο θα εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους πολίτες της Ένωσης. Γύρω τώρα για τις τοξικές ουσίες. σχετικά με τον ιατρικό εξοπλισμό. Οι εξοπλισμοί αυτοί δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν ε, τέτοιου είδους ε, ουσίες. Αυτό είναι ε, ο πρώτος κανόνας. Και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα αυτό και στην συνάντηση που θα κάνουμε τον μήνα Σεπτέμβριο για τον ιατρικό εξοπλισμό. Έχω χαθεί λίγο στις ερωτήσεις σας για τη διαφάνεια στον τομέα των κλινικών δοκιμών. Το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ε, την διάθεση πολλών πληροφοριών στο συστήματα ε, ελέγχου των προϊόντων. Στη συνάντηση της 8 η και 9ης Ιουλίου η Ιταλική Προεδρία κατέθεσε ένα σαφές αίτημα προς τα κράτη-μέλη να εκφράσουν την άποψή τους στην πληροφορική αυτή διαδικασία και να αξιολογήσουν την υποχρέωση του, κατασκευαστού, ε, του κατασκευαστή να ε, προσθέσει στην ενημέρωση του συστήματος περισσότερα στοιχεία ιδιαίτερα σε σχέση με τις, ε, με τις αρνητικές πλευρές της χρήσης ορισμένων ουσιών και τώρα θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τις απαντήσεις και οι απαντήσεις αυτές και τα δεδομένα γύρω από τις απαντήσεις αυτές θα είναι ελεύθερα δημόσια. Λοιπόν, ήταν τόσο πολλές ερωτήσεις που δεν τις ε, ελέγχω καλά. Τώρα, ο έλεγχος των αγορών. Κάποιες χώρες συμφωνούν, κάποιες άλλες ακόμα διαφωνούν στην δυνατότητα να προβλεφθεί ένας κεντρικός οργανισμός που θα είναι υπεύθυνος για τους μηχανισμούς ελέγχου, scrutiny mechanisms. Θα εκτιμήσουμε σε συνεργασία με τις άλλες χώρες την ανάγκη δημιουργίας ενός τέτοιου μηχανισμού, ιδιαίτερα για εξοπλισμούς υψηλού κινδύνου. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ τεχνικό, πολλά θέματα έχουν λυθεί Υπάρχουν άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε με επικοδομητικό πνεύμα και ελπίζω να καταλήξουμε σύντομα. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις, ευχαριστώ πολύ. Ναι πράγματι απαντήσατε σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις. Ξεκινάμε τώρα με το δεύτερο γύρο. Κόβατσεκ, ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Και εγώ Χαίρομαι γιατί η Ιταλική Προεδρία έβαλε την υγεία μέσα στις προτεραιότητες της, μίλησε για την πρόληψη, για την υγιεινή ζωή, το περιβάλλον, τη στρατηγική για τις χρόνιες ασθένειες, όλα αυτά πολύ σημαντικά. Υπάρχει όμως και το θέμα της άνησης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. πόλοι ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν πρόσβαση σε σωστή θεραπεία και διάγνωση. Αυτό μειώνει την, ε, το προσδόκιμο ζωής τους, τη διάρκεια της ζωής τους μάλλον. Η ανισότητα στις υγειονομικές υπηρεσίες προκαλεί περισσότερο η μετανάστευση. Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς και νοσοκόμας που φεύγουν από τις χώρες τους για να βρουν μια καλύτερη δουλειά αλλού. Αυτό είναι πρόκληση για ολόκληρη την Ένωση. Όλες οι χώρες της Ένωσης αφορούνται από αυτό το πρόβλημα. Ιδιαίτερα όμως τα καινούργια μέλη και αυτό φαίνεται από τις αναχώρασεις στάσεις του Συμβουλίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2014 και νομίζω ότι είναι αυτό μια καλή και σωστή βάση. Όπως είπε και ο συνάδελφος λέει για να κινητοποιηθούν τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι παραπάνω για να μεταρρυθμίσουν τις υγειονομικές τους υπηρεσίες. Η Κομισιόν το έχει δεχτεί ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον η Ιταλική Προεδρία θέλει να θίξει το θέμα των ανισοτήτων στο θέμα της περίθαλψης και δεύτερον τι σχεδιάζει να κάνει νομοθετικά ιδιαίτερα ως προς τα μέτρα διαφάνειας για τις τιμές των ιατρικών σκευαζημάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κόβατσεκ. Για τους σοσιαλιστές ο κύριος Παύλ Πότς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ένα πολύ απλό ερώτημα το οποίο συνδέεται με την αύξηση του επιπολασμού του καρκίνου και έχει να κάνει με τον ορισμό κριτηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδίως για τα αναφέρουμε στα κριτήρια που έχουν να κάνουν με την ανείχνευση των ενδοκρινικών διαταρακτών. Το πρόγραμμα της Ιταλικής Προεδρίας δεν είναι ιδιαίτερα σαφές σε ό,τι αφορά την ανείχνευσή τους. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που προτείνετε να αναπτύξετε τι κριτήρια θα δεχτείτε, ποια είναι τα σχέδιά σας στον τομέα αυτό. Ο Μπουζόη, κύριος Μπουζόη, έχει το λόγο. Θα μιλήσω αγγλικά. Κυρία Υπουργέ, η παρέμβασή μου που είναι σύντομη έχει να κάνει με ένα σημαντικό στοιχείο νομοθεσίας που είναι στο ψυγείο αυτή τη στιγμή, που είναι το νομοθέτημα για την ρύθμιση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων. Oh. Αναφέρομαι σε αυτό όχι μόνο γιατί ήμουν ο, ο συντάκτης γνωμοδότησης στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, αλλά γιατί έρχομαι από μια χώρα που ο κατάλογος των φαρμάκων που ε, αποζημιώνονται από τις ασφαλιστικές εταιρείε δεν έχει αλλάξει από το 2008. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν θα μπει σε αυτό το κατάλογο των φαρμάκων που ε, δίδεται επιστροφή στον ασθενή ή όχι. Υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες, αλλά τώρα αυτή η πρωτοβουλία έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση της Ιταλικής Προεδρίας για το θέμα αυτό και αν είναι θετική η γνώμη της Ιταλικής Προεδρίας θα ήθελα να ζητήσω να ξεμπλοκάρετε τη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας και λυπάμαι πάρα πολύ που σύντομα πρέπει να πάρει στο αεροδρόμιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια κύριε Υπουργέ για την πλήρη απάντησή σας και για τις ενθαρρυντικές απαντήσεις που δώσατε στους συναδέλφους. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τους κινδύνους οι οποίοι δημιουργούνται από το Wi-Fi. Κάποιες δημοσιογραφικές πηγές, όλο ένα και πιο ισχυρές, ε, αρχίζουν να διαδίδουν ότι η έκθεση σε χαμηλού ε, επίπεδου ε, φάσματα συχνοτήτων μπορεί να είναι επικίνδυνες για την υγεία και ότι υπάρχει ένα έγγραφο 350 σελίδων το οποίο λέγεται Διεθνές ε, Συμπόσιο Συμπόσιο 05-6904, μέσω του οποίου η Διεθνής Οργάνωση Υγείας ε, ε, βλέπει ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας λόγω της έκθεσης σε Wi-Fi. Ε, καταλαβαίνετε ότι η υγεία είναι μια προτεραιότητα για, για τα εξάμεινα και το συγκεκριμένο της Ιταλικής Προεδρίας για την πρόληψη ασθενειών όπως ο καρκίνος, ε, τα καρδιαγγειακά και τα αναπνευστικά. Ε, εσείς έχετε υπόψη σας τα δεδομένα αυτά θα τα αντιμετωπίσετε και τι πρωτοβουλίες σκοπεύετε να πάρετε για να προστατεύσετε την υγεία των πολιτών σε όλα τα κράτη-μέλη λόγω ακριβώς αυτών των προβλημάτων. Ένα άλλο ερώτημα που θα αναθέσω αφορά τον μητρό των όγκων. Ε, η Ιταλική Προεδρία πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει μια ομογενοποίηση των μητρών σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό στοιχείο πρόληψης αν κάτι τέτοιο υπάρξει. Φαρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλημέρα σας κυρία Υπουργέ και σας συγχαίρω για την παρέμβασή σας. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει προβλήματα για τη δημόσια υγεία, ιδίω στι χώρε που έχουν πληγεί από αυτή την κρίση, ιδίω στη δική μου χώρα, την Πορτογαλία. Υπήρξε μία αύξηση στις μεταδοτικές ασθένειες και αναφερθήκατε στο θέμα των ψυχικών ασθενειών λόγω του στρες που ήταν πηγή και θανάτων. Οι δείκτες μας για τις ψυχικές ασθένειες όπως είναι η κατάθλιψη και οι αυτοκτονίες, ιδίως στις πιο τροτές κοινωνικές τάξεις έχουν αυξηθεί. Συγχρόνως, για λόγους οικονομικούς έχει μειωθεί η περίθαλψη σε όλες τις χώρες οι, τα τέλη που καταβάλουν οι χρήστες των εθνικών υπηρεσιών υγείας αυξήθηκαν πάρα πολύ και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν όλο και μεγαλύτερες ανισότητες στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Πώς βλέπετε κυρία Υπουργέ το ρόλο της Ιταλικής Προεδρίας για να αντιμετωπιστούν αυτές οι αλλαγές. Θα πάρετε συγκεκριμένη δράση βάσει της αρχής της επικορικότητας για να υπάρξει μεταλαμβάνευση βελτίστων των πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών για την καλύτερη χρησιμοποίηση και λειτουργία των υγειονομικών τους υπηρεσιών και για την πρόληψη των ασθενείων. Και όπως είπατε, η υγεία των πολιτών μας είναι αδιαπραγματεύτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρντίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη γιατί έχουμε πράγματι πει πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ την Υπουργό για την συνάντηση αυτή. Νομίζω ότι η στάση την οποία παρουσίασε είναι συμβατή. με την έκθεση της Υπηρεσίας για την Ευρώπη της Διεθνούς Οργάνωσης Υγείας για τις μη μεταδοτικές ασθένειες. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα σε πάρα πολλές χώρες. Πράγματι η πρόληψη είναι κάτι το οποίο απαιτείται για να αποφύγουμε την διάδοση των ασθενειών αυτών που οδηγούν σε πολλές απώλειες ζωής. Σημερίζομαι λοιπόν τις απόψεις σας, θα ήθελα να μάθω αν είναι μία από τις προτεραιότητάς σας. στην Αλμπουφέιρα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είχε παρουσιάσει ένα κατάλογο προτεραιοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα θέμα το οποίο, στο οποίο επιμένει η οδηγία για την διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της φροντίδας των ασθενών. Είναι κάτι το οποίο ανοίγει δρόμους για το μέλλον Υπάρχει από τη μία ανάγκη για την εξορθολογιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα επιτρέψουν να υπάρχουν και εξοικονομήσεις ποσών σε μικρές χώρες που δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν ειδικά κέντρα σαν παράδειγμα για σπάνιες ασθένειες και γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε τι θα συζητήσετε στο Μιλάνο όταν τεθούν τα θέματα της υγείας και πώς μπορείτε να συνεργαστείτε με τα μέλη του Κοινοβουλίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, έτσι ώστε να προωθηθεί η οδηγία αυτή τόσο χρήσιμη για το Κοινοβούλιο και τους πολίτες. Ίσως θα μου άρεσε βέβαια η χώρα μου να είναι αυτή η οποία θα δώσει περιθώρια για την υιοθέτηση και την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κινήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Υπουργό για την προσεκτική και λεπτομερή παρουσίαση του προγράμματος της στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ε, την ευχαριστώ για, ε, ε, για την ακρίβεια σε αυτά τα οποία μας είπε. Έχω μία ερώτηση την οποία θα ήθελα να θέσω πάνω σε ένα θέμα στο οποίο έχετε ήδη αναφερθεί αρχικά τον Απρίλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκλεισε την πρώτη του ανάγνωση για, την, ε, για τον έλεγχο των ε, τροφίμων. Ένα θέμα περίπλοκο αλλά και πολύ σημαντικό έτσι ώστε να υπάρξουν εγγυήσει ε, για την προστασία των τροφίμων μας. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν τι πρωτοβουλίες σκοπεύετε να αναλάβετε σε έναν τομέα στον οποίο το Συμβούλιο από ό,τι φαίνεται δεν έχει κάνει μέχρι τώρα πολλά. Και πώς μπορείτε να βοηθήσετε έτσι ώστε να βελτιωθούν οι έλεγχοι στην τροφιμική αλυσίδα, σύμφωνα με συγκεκριμένους κατελάχιστον αποδεκτούς κανόνες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης έχει ζητήσει να υπάρξουν ε, ενημερωμένα και από κοινού δεκτά συστήματα εκπομπής συχνοτήτων. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην πολιτική λιτότητας που δεν έχουν φυστεί ούτε των υπηρεσιών υγείας για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και θα ήθελα να αναφερθώ στις στατιστικές μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα στην υγειονομική περιθέλψη, όλο και πιο μεγάλο μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών περιοχών της Ευρωπαϊκής Υπήρου κυρίως αυτών που έχουν πληγεί από την κρίση. Η κατάσταση στην Ιταλία έχει δει πολλές περιπτώσεις που έχουν ε, καταρρεύσει οι υπηρεσίε υγεία ουσιαστικά έχουν στραφεί προ την αναζήτηση του κέντρου και έχουν αντικαταστήσει τι δημόσιε υπηρεσίε. Είναι μια κατάσταση στην οποία ο ασθενή γίνεται πελάτη. Η υγεία γίνεται ένα αντικείμενο εμπορία. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβετε υπόψη τις αποδοχές των ε, ε, διοικητών των νοσοκομείων και των πολιτικών που είναι και μια από τις πηγές της τωρινής κατάστασης και της κρίσης και που οδηγούν στην υπονόμευση της υγείας των πολιτών. Κάτι το οποίο προστατεύει και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να σας υπενθυμίσω επίσης την ε, πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών που θέλει να σταματήσουν τα πειράματα σε ζώντα ζώα και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση της Ιταλικής Προεδρίας για τα πειράματα σε ζώντα ζώα. Άλλοι δύο μιλητές, η κυρία Ιούσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την κυρία Υπουργό. Εγώ ήθελα να σας θέσω και μία και να σας μεταφέρω τα σχόλια της κυρίας Γκροστέτη η οποία δεν μπορούσε να τα παρούσε και έλεγε ότι έχουμε περάσει τα πρώτα πέντε χρόνια σε σχέση με την ε, εφαρμογή μιας οδηγίας για τα φαρμακευτικά σκευάσματα στην Ευρώπη, αλλά οι διαδικασίες επί παραβάση δείχνουν ότι η νομοθεσία αυτή δεν τηρείται από τα κράτη-μέλη. Παραγωγός χάρη στη Γαλλία και την Ιταλία έχουν ε, μεταγραφεί όλα αυτά στην εθνική νομοθεσία ώστε να υπάρχει δυνατότητα να τίθενται εκτός εμπορίας όλα ορισμένα φάρμακα. Και υπήρξαν ρυθμίσει που έγιναν μόνο για λόγου προπολογισμού παρά το γεγονό ότι υπάρχουν φάρμακα αναλλακτικά τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι ασθενεί στη Γαλλία και την Ιταλία. Όλα αυτά είναι ένα επικίνδυνο προηγούμενο <clears throat> και σημαίνουν μια πραγματική πρόκληση για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα φάρμακα κυκλοφορούν για συγκεκριμένες ε, ενδείξεις και μόνο και συμπτώματα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους λόγους. το να παραγνωρίζονται αυτές οι ενδείξεις για την κυκλοφορία των φαρμάκων είναι κάτι το οποίο μπορεί να θίξει την υγεία των ασθενών γιατί στις περιπτώσεις αυτές δεν τηρούνται τα πρότυπα για τα οποία έχουν εγκριθεί τα αντίστοιχα αυτά φάρμακα. Αυτή η παράβαση λοιπόν των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κράτη-μέλη ουσιαστικά υποσκάπτει τη βάση της ρύθμισης των φαρμακευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μειώνει την πρόσβαση των ασθενών σε συγκεκριμένα φάρμακα, κυρίως μειώνει και τις δυνατότητες να υπάρξει καινοτομία και περαιτέρω έρευνα για τα θέματα αυτά. Το ερώτημα μου είναι αν έχει σκεφτεί η Ιταλική Προεδρία να εξασφαλίσει την προστασία του κοινωνικού κεκτημένου και να το κάνει προτεραιότητά της και αν η Κομισιόν είναι έτοιμη να εφαρμόσει μια πιο <clears throat> αυστηρή πολιτική στην περίπτωση που παραβιάζεται αυτή η νομοθεσία για τα φαρμακευτικά από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ την κυρία Ιούζο. Τελευταία παρέμβαση είναι από τον Άλτο Πατρισέλο και μετά θα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την παρουσίασή σας. Συμφωνώ στην ανάγκη να δημιουργηθεί μια στρατηγική εναρμονισμένης πρόληψης στις διάφορες χώρες. Θα ήθελα να ζητήσω το εξής, ε, κυρία Υπουργέ. Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να ενισχύσετε την ευρωπαϊκή πλατφόρμα γύρω από τις λεγόμενες σπάνιες ασθένειες, των οποίων το κοινωνικό κόστος, παρότι αφορά ένα μικρό αριθμό πολιτών, είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε δημοσιονομικό επίπεδο. Μια άλλη ερώτηση η οποία αφορά τη χώρα μου κυρίως. Ε, σκοπεύετε εσείς να επανεξετάσετε τις ιδιαίτερα περιοριστικές διατάξεις στην Ιταλία για τα πειράματα στα ζώα. Στην Ιταλία οι έρευνες ε, είναι πάρα πολύ δύσκολες ε, και και αναφέρομαι όχι σε μεγάλα ζώα αλλά σε αρωραίους και σε ποντικούς κυρίως. Και δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τις διάφορες κατηγορίες ζώων που χρησιμοποιούνται στην εργαστηριακή έρευνα. Ιδιαίτερα στα πλαίσια της μάχης που δίνουν τα φαρμακευτικά εργαστήρια και βιομηχανίες στον τομέα της έρευνας είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Ένα άλλο θέμα, και επανέρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία Γκαρντίνη, είναι η διασύνοριακή φροντίδα για τους ασθενείς. Αν υπάρχει δυνατότητα να εργαστούμε στον τομέα της ενιαίας τιμολόγησης έτσι ώστε να αποφύγουμε καταχρήσεις. Ευχαριστώ Άλντο. Δεν έχουν ζητήσει άλλοι τον λόγο. Έχουμε εξαντλήσει πλέον όλα τα αιτήματα, ε, τις ερωτήσεις μάλλον και θα δώσω το λόγο στην Υπουργό ε, για να μπορέσει να δώσει, αν είναι δυνατόν βέβαια, απαντήσεις στις ερωτήσεις οι οποίες έχουν τεθεί. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Είναι θέματα τα οποία θα λάβουμε υπόψη μας και σαν κράτος μέλος αλλά φυσικά και σαν Προεδρία. Θα ξεκινήσω από το θέμα της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της υγείας. Στην Ιταλία έχουμε μόλις εγκρίνει και θέσει εφαρμογή την οδηγία για τη διασυνοριακή συνεργασία. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για μας ιδιαίτερα για την ίδια την Ευρώπη. Αν σκεφτείτε κάπως προσεκτικά η οδηγία αυτή είναι η πρώτη οδηγία η οποία ασχολείται με τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τους πολίτες, με τα δικαιώματά τους, όχι μόνο τα δικαιώματα τα οικονομικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και όπως όλες οι οδηγίες βέβαια, οι οποίες ξεκινούν με πάρα πολλές καινοτόμες ε, απόψεις, ε, υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστούν σωστά. Η οδηγία στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται από τα διάφορα κράτη-μέλη περιλαμβάνει για να χρησιμοποιήσω ένα ιατρικό όρο αντισώματα. Αντισώματα έτσι ώστε να μην χρησιμοποιηθεί σαν μέσο υγειονομικού τουρισμού και καταχρήσεων. Αντίθετα έχει όμως πολλά καινοτόμα στοιχεία φανταστείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν έναν μεγάλο χώρο στον οποίο ε, μπορούν να γίνουν δοκιμές σε σχέση με τις σπάνιες ασθένειες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη να συγκεντρώσουμε ε, τα κέντρα έρευνα σε εθνικό επίπεδο και σε ορισμένες περιπτώσεις δοκιμών εργαστηριακών το εθνικό επίπεδο δεν αρκεί και το ευρωπαϊκό ή το διεθνές είναι απαραίτητο. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια ανάγκη ανάπτυξης και απόδοσης εγγυήσεων για τους πολίτες έτσι ώστε να μπορέσουν να θεραπευθούν με τον σωστό τρόπο. Και επίσης έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε και διάφορα προβλήματα ανταγωνισμού στον τομέα της τιμολόγησης των προϊόντων υγείας. Εμείς το Νοέμβριο θα οργανώσουμε ένα σημαντικό, ελπίζω, μια σημαντική συνάντηση για το θέμα αυτό στη Βενετία. Δεν μπορούσα να το κάνω στο Μιλάνο. Θα γίνει λοιπόν στη Βενετία αυτή η συνάντηση και θα πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος στην συνάντηση αυτή και με τα μέλη του Συμβουλίου και με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συζητήσουμε τις δυνατότητες που έχει η οδηγία αυτή και για την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας αυτής στον υπόλοιπο κόσμο, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα αντιμετωπίσουμε και πιο συγκεκριμένα το θέμα των ογκολογικών προβλημάτων και μέσω της πρόληψης, της φροντίδας και της καινοτομίας στα πλαίσια της διασυνοριακής ε, οδηγίας. Πάντα για την πρόληψη των όγκων ε, μου τέθηκε μία ερώτηση την οποία δεν βρίσκω. Λοιπόν, μου τέθηκε μία ερώτηση ε, στην αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιπροσωπεύουν οι όγκοι στην Ευρώπη σε σχέση με τις στρατηγικές ε, που θα εφαρμοστούν στο μέλλον και πώς θα αξιολογηθούν ε, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί ήδη. Ε, όπως είπαμε, οι τρόποι ζωής μπορούν μέσω της σωστής, όταν ακολουθούνται σωστά, με μειωμένο αλάτι, με μειωμένο αλκοόλ, με μειωμένο λίπος και με σωστή άσκηση θα εξασφαλίσουμε πάρα πολλές βελτιώσεις. Επίσης λοιπόν θα προωθήσουμε την ζωή, η μια, ένα τρόπο ζωής ο οποίος θα πρέπει να είναι συμβατός με την υγεία, όχι μόνο σε επίπεδο θεραπευτικό, γιατί γνωρίζετε ότι υπάρχουν προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης και στην πρόσβαση των πολετών ε, στα μέτρα διάγνωσης και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Και υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε επίσης και κάποιες εκστρατείες για την μεγαλύτερη ακόμα χρήση των μεθόδων εμβολιασμού για τα θέματα της αηφορίας και της καινοτομίας. Να πω ότι η καινοτομία δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυστηρά οικονομικό. Είναι κάτι το οποίο άπτεται του συστήματος υγείας βέβαια, άπτεται όμως και της ικανότητας των χωρών να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις τεχνολογικές καινοτομίες. Εμείς κατά τη διάρκεια της ανεπίσημης συνάντησης θα ασχοληθούμε και με το θέμα αυτό το οποίο είναι κρίσιμο για τις πολιτικές υγείας των χωρών μας στο μέλλον. Πρόκειται για ένα θέμα κρίσιμο και για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Και όπως φαίνεται στα πλαίσια του συστήματος για την υγεία υπάρχουν και άλλοι τομείς της ανάπτυξης και της έρευνας που συνδέονται η οικονομική κρίση εκτός από το να περιορίζει ε, ε, τις ε, προσβάσεις στη διάγνωση και στη θεραπεία μερικές φορές μειώνει και τις ικανότητες στον τομέα της έρευνας. Στην άτυπη συνάντηση λοιπόν αυτά θα συζητήσουμε. Ποιες είναι οι διαθέσιμες στρατηγικές για να βελτιώσουμε την καινοτομία στα ερευνητικά μας συστήματα έτσι ώστε να εγγυηθούμε στους συμπολίτε μας τις μέγιστες επιδόσεις στον τομέα της, στον τομέα της υγείας. Η Ευρώπη πάντα έδωσε στους συμπολίτε μας έδωσε εγγυήσει στους συμπολίτε ε, για την πρόσβαση στις καλύτερες ε, δυνατές ε, φροντίδες υγείας, στον τομέα της υγείας. Χρησιμοποιήσαμε στο μέγιστο βαθμό την τεχνολογική ε, καινοτομία, έχουμε ένα υψηλό επίπεδο, ε, ε, υψηλό επίπεδο και σε πολιτιστικό, στον πολιτιστικό τομέα και στον τομέα τον οικονομικό όμως σε σχέση με άλλες χώρες όπως η ΕΠΑ και η BRICS. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια διαφορετική μορφή πρόσβαση στην κοινοτομία και αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου. Η Ιταλική Προεδρία επίσης προετοίμασε το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με συνεργασία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν μια πολύ χρήσιμη συνεργασία. Διατυπώσαμε ένα έγγραφο το οποίο θα τονώσει την ανάπτυξη, θα διευκολύνει συγγνώμη, την ανάπτυξη, θα διευκολύνει την έρευνα για φαρμακευτικές ουσίες και προϊόντα, που θα καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών και σε επίπεδο νέων ε, πολλά υποσχόμενων θεραπείων. Ένα άλλο θέμα το οποίο τέθηκε αφορά την διαφάνεια, την οδηγία για την διαφάνεια και για την τιμολόγηση της φροντίδας στον τομέα της υγείας. Είναι σημαντική οδηγία η οποία ορίζει επίπεδα διαδικαστικού τύπου για να υπάρχουν εγγυήσεις στον τομέα της λήψης αποφάσεων σχετικά με το κόστος της φροντίδας της ιατρικής και της επιστροφής του κόστους. Ε, υπάρχουν και κάποια στοιχεία στις οδηγίες αυτές τα οποία, ε, στα οποία υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς και υπό το φως των αποτελεσμάτων της τελευταίας συνάντησης της ομάδας εργασίας ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Περιμένουμε τις τελικές θέσεις ε, από πλευράς των κρατών μελών έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε τις πιθανές αντιτιθέμενες απόψεις και να μπορέσουμε να προτείνουμε μια ε, λύση αντικειμενική και αποδεκτή. Τώρα, σχετικά με τις προτάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, εφόσον συγκεντρωθούν οι προϋποθέσεις θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε. Ε, η συγκυρία είναι κρίσιμη σχετικά με την διαδικασία καθορισμού των τιμών για την επιστροφή του κόστους των φαρμάκων. Ε, ιδιαίτερα στα φάρμακα για την υπατήτηδα γάμα. Θα πρέπει να πω εδώ ότι αναλύουμε το συγκεκριμένο θέμα το κάνουμε προσεκτικά με τα κράτη-μέλη και υπό το φως των νέων κρίσιμων καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση η οποία να γίνεται αποδεκτή από όλους. Για το ερώτημα το οποίο έχει τεθεί για τα πειράματα σε ζώα. Οι προβλέψεις ε, ζητούν να μην ε, υπάρχει δυνατότητα, περιλαμβάνεται η πρόταση να σταματήσουν τα πειράματα σε ζώα ή να προβλεφθεί η ελάχιστη δυνατή θεσία των ε, ζώων μέσω της κατανομής και της αποκοινού τέλεσης των πειραμάτων σε ζώα για να μειωθεί ο αριθμός τους. Ναι. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό. Για για την ερώτηση για τα, για τα γενώσιμα. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να παρακολουθήσουμε σωστά τους κανόνες και την εφαρμογή τους γιατί πάνω από οτιδήποτε άλλο υπάρχει η ασφάλεια του πολίτη, του ασθενούς και σε σχέση με την Προεδρία και σε σχέση ε, ε, μου προσωπικά ως Υπουργού. Φυσικά τα κράτη-μέλη με επικουρικό τρόπο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα off-label φάρμακα στο βαθμό που διασφαλίζουν την ασφάλειά τους και μπορεί να υπάρξουν και ε, διαδικασίες καινοτόμε οι οποίες θα οδηγήσουν στην χρήση αυτών των νέων σκευασμάτων. Λοιπόν, εμείς σαν Προεδρία νομίζω ότι δείχνουμε σε όλους ότι ε, στο κέντρο της πολιτικής μας για τα φάρμακα βρίσκεται η ασφάλεια του πολίτη. Ε, για την ερώτηση της κυρίας Κινίση. Στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων ε, και στον έλεγχο φυσικά όλης της διαδικασίας της παραγωγής τροφίμων απαιτείται να υπάρχει μια σωστή νομοθετική ρύθμιση με τα κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας. Αυτό όμως ε, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με κοινοτικούς κανόνες ελέγχου που θα ε, ε, αξιολογούν τον κίνδυνο. Είναι απαραίτητο λοιπόν όλες οι χώρες για να αποφύγουμε στο μέλλον στρεβλώσεις να κάνουν τον ίδιο, με τον ίδιο τρόπο ότι τον έλεγχο τον οποίο καλούνται να κάνουν. Θα αναζητήσουμε τη συνένεση του Συμβουλίου στον τομέα αυτό, γιατί σήμερα υπάρχουν διιστάμενες απόψεις, αλλά νομίζω ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, για το οποίο όλοι ενδιαφέρονται, και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα εναρμονίσουμε τις αποκλίνουσες θέσεις. Τελείωσα. Τελείωσα λέει υπουργό. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό Λορεντσίν, την Προεδρεύουσα λοιπόν του Συμβουλίου για την ε, διαθεσιμότητά της, γιατί απάντησε σε, ε, σε, ένα τεράστιο αριθμό ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ όλους. Κλείνει η συνεδρίαση της Επιτροπής. Αύριο έχουμε τις, τους συντονιστές και στις 3 Σεπτεμβρίου θα έχουμε την νέα μας μορφή, ε, τη νέα μας συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ.